Okay. Are you ready? Είστε έτοιμοι? Μυστική ψηφοφορία λοιπόν είπαμε. Αρχίζουμε με την κυρία Έντιν Μπάουερ. Ψηφίστε παρακαλώ. Ωραία. 40 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Συνεχίζουμε. Αλεχάνδρο Σέρκας. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote Τέλος της ψηφοφορίας. Πάλι δυνατό το αποτέλεσμα, 40 υπέρ, 1 κατά. Και Jean-François Mezier τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote. Πέρας της 38 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 2 αποχές. Αυτό σημαίνει ότι εκλέγονται και οι τρεις υποψήφοι. Οπότε θα συστηθούν από μας για ορισμό. Δύο είναι. Ήτανε μάλλον χτες το απόγευμα εδώ στην Επιτροπή μας. Θα σταλεί λοιπόν ο κατάλογο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε ω κοινοβούλιο στα επόμενα βήματα τη διαδικασία, δηλαδή την έγκριση από τη διάσκεψη των προέδρων και τον ορισμό τους από τον πρόεδρό μα. Ευχαριστούμε και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία τώρα που αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βάσει του άρθρου 53 θεωρώ, όσο έχω το δικαίωμα βάσει του άρθρου αυτού, ότι κάποιες τροπολογίες δεν είναι παραδεκτές επειδή δεν έχουν να κάνουν με τις αμμοδιότητες της Επιτροπής μας. Πρόκειται για τις τροπολογίες 3, 10, 11, 14, 22, 30, 31, 36 και 48. Οπότε οι συντάκτες τους, αν θέλουν να τις επανακαταθέσουν, να τις επανακαταθέσουν απευθείας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. προθεσμία είναι 31η Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι. Παρακαλώ κύριε Μακιντάιρ. Πρόεδρε, με εκπλήσει ο τρόπος που χειρίζεστε αυτό το θέμα γιατί πρόκειται ακριβώς για τις ίδιες τροπολογίες που κατατέθηκαν με την έκθεση Πυρίνσκι για τέτοια ακριβώς θέματα. Τότε δεν εκφράσατε καμία ένσταση. δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο λόγος είναι ότι οι τροπολογίες αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή Προπολογισμών. Αυτός είναι ο λόγος. Και είναι κάτι που συζητήθηκε σε βάθος πριν ληφθεί η απόφαση αυτή. Καλώς. Οπότε όσοι θέλουν μπορούν να τις επανακαταθέσουν απευθεία στην Επιτροπή Προεπολογισμών. Και η προθεσμία είναι 31η Ιανουαρίου, όπως σας είπα. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα και αρχίζουμε με την τροπολογία αριθμός 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 8 λοιπόν. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 είναι από τις μη αποδεκτές. Η 11 επίσης. Τροπολογία 12 υπέρ κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Α, από το ψήφισαν ένας παραπάνω. Ωραία, εγκρίθηκε 24 ψήφοι υπέρ. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 μη αποδεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε με 27 υπέρ.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Δεύτερο τμήμα. Γιατί το πρώτο καταπίπτει. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 26 ψήφι κατά. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 δεν είναι αποδεκτή. 31 δεν είναι αποδεκτή. 32 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. μη αποδεκτή. 37 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 42 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για τη 42. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 44. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική C γάμα. Α, όχι, προηγουμένως θα ελέγξουμε για τη 44 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 26 υπέρ εγκρίθηκε. Τώρα συμβαστική C γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 46. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε με 23. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 Α, θέλετε να ελέγξουμε για τις 47. Ωραία. Ηλεκτρονικά λοιπόν. 47 ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Με 27 ψήφους υπέρ. 48. μη αποδεκτή. 49 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 54. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίθηκε 37 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 59 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική FB. Σίγμα ταφ Β. Μπορούμε να έχουμε ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. ήταν οι σοσιαλιστές. Καλώς. Ωραία, για τη συμβαστική λοιπόν σίγμα τάφ β, FB. Έτσι, για αυτήν θέλετε ονομαστική, σωστά. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι για να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 59 ή τη συμβαστική F, τη συμβιβαστική FB, συμβαστική σίγμα τάφ β. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε Α, πρέπει 11 να σηκωθούν για να το ζητήσουν. 11. Ωραία. Είναι αρκετή. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία για τη συμβαστική FB. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας και απορρίφθηκε με 27 ψήφους κατά. Τροπολογία 62, δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, λέω. 63, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 63. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 50. Διακόπτη πρόεδρος. 64, 65 και 66 καταπίπτουν. Οπότε πάμε στην τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 66. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ. 60 7 πίπτη και 68. Συμβαστική H ή τα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I για τα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69. πίπτη Και η 71 υπέρ. Α, όχι διορθώνει ο πρόεδρος, λάθος. Και 71 καταπίπτει. Πάμε στην τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 72. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 27 ψήφους κατά. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία Δύο θεωρείται εγκεκριμένη. Οπότε δεν την ψηφίσουμε. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 καταπίπτει. Αυτά. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία απαλλαγών. Ξεκινάμε το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Α, συγγνώμη, 9 διορθώνει πρόεδρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 13. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε τη 17. Πέρες και απορρίφθηκε με τρεις ψήφους διαφορά. 19 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σχέδιο γνωμοδότησης τώρα, το τροποποιημένο, παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 39 ψήφοι υπέρ, 8 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συνεχίζουμε τώρα. Και περνάμε στο ETF, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική Εκπαίδευση, απαλλαγή για το έτος 2016. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση συνολικά όπως τροποποιήθηκε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας, 41 προς 6. 6 ψήφι, 3 αποχές. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και προχωρούμε. Προϋπολογισμός εκτέλεση των προπολογισμών των ευρωπαϊκών οργανισμών για το δημοσιονομικό έτος. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και μετά το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται 39 προς 6. Τέσσερις αποχές.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 5, συμβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για να ψηφίσουμε για την 16. Πέρα στις ψηφοφορίες για τη 16. Εγκρίνεται 37 προς 12. Αλλά να σηκώνετε τα χέρια σα έτσι κι αλλιώ. Και μετά ψηφίζουμε το σχέδιο δογματοδότησης ω τροποποιήθηκε. Υπέρ. Είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία, ναι, με συγχωρείτε. Πέρα. Εγκρίνεται με 42 ψήφου υπέρ. 8 κατά. Καμία εποχή. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Και μετά περνάμε στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ανία ψηφοφορία. Μάλλον μία μόνο ψηφοφορία για την πρώτη απολογία. Υπέρ, κατά. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την πρώτη τροπολογία για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Καμιά φορά πρέπει να έχει κανεί πολύ ξεκάθαρες οδηγίες, έτσι κύριε Κάζα. Αλλά αυτή τη φορά ήσασταν στο στρατοπεδό που κέρδισε, 28. Ψήφι και 22 αποχές. Μετά ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση ω τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία και αυτή άρχεται. Πέρας. 42 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Πάμε στην Όσα. Παράγραφος 2, πρώτη τροπολογία, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο, μάλλον τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και μετά ψηφίζουμε το σχέδιο γνωματοδότησης ως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται 42 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Και καμία αποχή. Ευχαριστούμε και τώρα απαλλαγή. Σχέδιο οικονομοδότησης για την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης της κυρίας Μπόιλαν. Τροπολογία πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές να ε, ελέγξουμε για την συμβαστική εννέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. 38 ψηφί, υπέρ, 8 κατά, 2 εποχές. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά να ελέγξουμε για την τροπολογία 26 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 27 προς 22 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ Κατά. Α, 31, να κάνουμε έλεγχο. Επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο ψεύτια χώρα. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Δυστυχώς. Δύο. Συμβαστική δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά να κάνουμε επαλήθευση για την 45, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά να κάνουμε έλεγχο για την 57 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 28 προς 22 θετικές ψήφους 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά έλεγχος για την 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τι γίνεται. Α, απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 η επόμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έλεγχο για την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και αυτή. 76 Πρώτο τμήμα. Όπως ζήτησαν οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Αγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να κάνουμε έλεγχο για την 86 λοιπόν. Πέρας. Απορρίφθηκε. 28 ψήφι κατά. Προς 21. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 8 υπέρ. Κατά. Να κάνουμε παλήθευση για την αιτιολογική και την ε, τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία και τώρα έλεξε. Απορρίφθηκε. Τέσσερις ψήφι διαφορά. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε, αλλά να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία. Άρχεται, έρχεται Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία, έλεξη ψηφοφορία, εγκρίνεται με 42 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 5 αποχές. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια την κυρία Μπόιλαν. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι απαιτήσει επιβολής και ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, το οποίο αποτελεί και σημαντικό μέρος της, του κανονισμού μάλλον, τον οποίο επεξεργαζόμαστε, περί αποσπάσεως εργαζομένων. Όταν θα υπάρχει κάποια ησυχία στην αίθουσα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή αλλά να σας δώσω ακόμη ένα λεπτό για να μπορέσετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα και να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια κυρία Λαντζόβα. Κοιτάξτε, βεβαίως δεν είναι και τόσο ευχάριστο να αρχίζω να ομιλώ όταν Όλοι βρίσκονται στην φάση της αποχωρήσεως. Βεβαίως μετρά η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Δεν είναι εύκολη η συζήτηση σήμερα και θα ήθελα να ακούσω από εσά τις διαφορετικές απόψεις γιατί νομίζω ότι η συζήτηση θα διαμορφωθεί ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα όμως πρώτα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταθέτει την πρόταση για την απόσπαση των οδηγών μέσα στο μεγάλο αυτό ε, πακέτο μέτρων για ε, την απόσπαση εργαζομένων. Επειδή είμαι εισηγήτρια αλλά και σκιώδη εισηγήτρια για την απόσπαση εργαζομένων, νομίζω ότι είναι σαφέ ότι οι οδικέ μεταφορέ χρειάζονται ειδικά τομεακά μέτρα. Ο τομέα λοιπόν των μεταφορών είναι πολύ ειδικό και άρα χρειάζεται ειδικέ ρυθμίσει. Κανόνε που να είναι ξεκάθαροι, ενιαίοι και εύκολο να εφαρμοστούν για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και βεβαίως η απασχόληση των προσώπων στον κλάδο αυτό. Όπως συμπεραίνει η μελέτη αντικτύπου, οι διάφορες απαιτήσει δεν αποδίδουν τον πολύ κινητικό κόσμο των οδηγών και αυτό επιβάλλει ιδιαίτερο ε, διοικητικό βάρος στους επιχειρηματίες και δυσχεραίνει τις διαμεθοριακές συναλλαγές. Στο σχέδιο γνωμοδοτήσεώς μου κάνω μια προσπάθεια να διευκρινίσω και να απλουστεύσω τους κανόνες. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο προτεραιότητές μου κατά την σύνταξη της ε, γνωμοδοτήσεως. Στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως λοιπόν τονίζω πρώτα ότι δεν περιλαμβάνω το transit, την διαμετακόμιση. Απλώς για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, διότι η διαμετακόμιση εν πάση περιπτώσει δεν θεωρείται ως κατάσταση απόσπασης ε, οδηγού. Επίσης, απομακρύνομαι από την καταμέτρηση των ημερών ε, για τις διεθνείς μεταφορές όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι εμένα με απασχολούν οι κανόνες που συζητούνται ακόμα στην γενική οδηγία απόσπασης και ιδίως ό,τι αφορά τις αμοιβέ, συλλογικές συμβάσεις, την μακροπρόθεσμη απόσπαση και ούτω καθεξής. Αυτά ακόμη είναι ανοιχτά και ασαφή. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν πού θα καταλήξουν μέχρι ότου καταλήξουν οι διαπραγματεύσει στον τριμερή διάλογο. Γι' αυτό δεν είναι ρεαλιστικό να εφαρμόσουμε του ίδιου κανόνε που αρχικώ προορίζονται, α πούμε, για τον τομέα τη οικοδομή στι μεταφορέ. Διότι οι οδηγοί μπορεί τελικώ να καταλήξουν να εργάζονται σε διαφορετικέ χώρε και μέσα σε μία ημέρα. Θα είναι λοιπόν τεράστιο διοικητικό βάρο να εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνε απόσπαση στου οδηγού, μεταξύ αυτών και να υπολογίζονται οι αμοιβέ και η ακρίβειά τους. Δεύτερο, ό,τι αφορά το λεγόμενο καμποτάζ. Συμφωνώ γενικά με την επιβολή ορισμένων στοιχείων από την οδηγία απόσπασης. Θα τα βρείτε αυτά και στο σχέδιό μου. Τέλος, βλέπω κάποια προβλήματα μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης των ημερομηνιών θέσης εφαρμογή ανάμεσα στην αναθεωρημένη ε, οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και του ειδικότερου νόμου λέξη σπετσιάλη. Αυτό μου φαίνεται ότι χρειάζεται να επιληθεί. Γι' αυτό προτείνω να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά με ειδικότερη νομοθεσία έτσι ώστε να μην προκύψει σύγχυση. Επειδή όμως δεν υπάρχει σαφήνεια για τους κανόνες, ε, ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει ακόμη να εξαιρείται από την Γενική Οδηγία περί απόσπασης. Αυτά τα λέω για να εξηγήσω πώς ήθελα να είναι απολύτως απλό και σαφές το πρώτο σχέδιο. Βεβαίως και αναμένω να ακούσω τις ε, προτάσεις σας. Και οι τρεις φάκελοι που θα συζητήσουμε σήμερα είναι αλληλοσυνδεδεμένοι. Έχουμε λοιπόν ε, ας πούμε πολλά μέτωπα όπου εργαζόμαστε και γι' αυτό πρέπει να τα συντονίσουμε. Ολόκληρη η συζήτηση και για τους τρεις αυτούς φακέλους έχει ωστόσο κρίσιμο χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ η κυρία Γιασλοβιέτσκα δεν είναι σήμερα παρούσα. Την ε, αντικαθιστά ωστόσο η κυρία Κοσλόφσκα. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Κολλείεται δυστυχώ η συνάδελφό μου κυρία Γιασλοβιέτσκα. Έχει υποχρεώσει ανηλυμένε ήδη στην Πολωνία. Έχει όμω ε, το εξή σημείωμα το οποίο εγώ σα διαβάζω. Πρώτον, ευχαριστώ την Μαρτίνα για το θάρρος που έχει να ασχοληθεί με το δύσκολο αυτό θέμα, το οποίο είναι η εξέλιξη και η ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέα των μεταφορών είναι, έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα με, με πολύ έντονη κινητικότητα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ιδίω στον τομέα αυτό χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνε που είναι εύκολο να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν. Η εφαρμογή του δηλαδή. Χρειαζόμαστε κάποιε αρχέ που θα επιτρέψουν την ορθή λειτουργία του τομέα που θα αποτελέσει και την βάση βέβαια ή και αποτελεί ήδη την βάση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ασχολούμαι με θέματα αποσπάσεω εδώ και πολλά χρόνια και αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη υπόθεση. Η πλήρης εφαρμογή των αρχών που αρχικώ προβλέπονταν για του οικοδόμου, α πούμε, είναι αδύνατη στον τομέα των μεταφορών. Συμφωνώ λοιπόν με τη λογική που επικαλείται η εισηγήτρια και στην βάση τη οποία αποκλείει τι διεθνεί μεταφορέ από του κανόνε περί απόσπασης. Εκπροσωπώ την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θα αποδώσω εγώ ιδιαίτερη σημασία στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση οδηγών στις ε, διεθνείς μεταφορές, στην βάση αρχών που θα επιτρέπουν έντιμη και δίκαιη μεταχείριση όλων των απασχολουμένων για να μην καταλήξουν σε καταστάσεις όπου να ισχύουν για τον ίδιο οδηγό ταυτόχρονα πλοίων νομικά καθεστώτα. Νομίζω επίσης ότι η περίοδος των τριών ημερών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ βραχία, είναι πολύ περιορισμένη και δεν επαρκεί, διότι οι τρεις μέρες θα είναι τελικώ οι 18 ώρες εργασίας. Και νομίζω ότι οι μεταφορές δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τους κανόνες της μακροχρόνιας απόσπασης και γι' αυτό συμφωνώ με την εισηγητρία και σε αυτό. Κάποιες επιφυλάξεις έχουμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή όλων, δηλαδή και των περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων. Και μόνο στην Αυστρία οι σχετικές ε, ενώσεις έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 50 διαφορετικές ε, ταρίφες. Αυτό δεν θα διευκολύνει τους οδηγούς. Τα πράγματα αυτά θα πρέπει βέβαια να περιληφθούν στις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η έλεγχη για την εφαρμογή των κανόνων. Εδώ ευχαριστώ την Μαρτίνα για τις προτάσεις που κάνει, που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι υπέρ της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και για αυτό το λόγο η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών είναι απαραίτητη. Χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων σε ένα ενιαίο έντυπο. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατό να καταχωρούνται και να ε, ενημερώνονται τα δεδομένα το δυνατόν ταχύτερο. Σημαντικό είναι να γίνονται και έλεγχοι στους δρόμους. και να ελέγχονται και οι αμοιβέ, τα pay slip των εργαζόμενων σε αυτούς τους ελέγχους. Στη βάση του στήματο IMI που θα ενισχύσει και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Η θέση της ομάδας μου είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις τοποθετήσει. Το ζήτημα είναι δύσκολο και πολλοί από τους συναδέλφους με τους οποίους έχω συνομιλήσει μου τονίζουν τα προβλήματα των κατόνομα εταιριών, εταιριών χρηματοκιβωτίου που στην ουσία κρύβουν από πίσω τους αυτοαπασχολούμενους. Τα προβλήματα αυτά δεν πρόκειται να λυθούν εάν εφαρμόσουμε τους κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων ήδη από την πρώτη μέρα. Αντιθέτως, αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία θεών ζωνών. Χρειάζεται να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Ευχαριστώ πολύ η πρόεδρο. Σα ευχαριστώ και εγώ. Η σκιώδη. Α, είναι εδώ. Προσέρχεται, προσέρχεται. Ιδού αυτή. Μα πραγματικά ε, ήρθατε ακριβώ στη σωστή χρονική στιγμή κυρία Ρέγνερ. Σα αφήνω να ε, ανασάνετε μια στιγμή, να καθίσετε. Η κυρία Ρέγνερ, ευχαριστώ που ε, με περιμένατε, ήρθα πράγματι με λίγη καθυστέρηση. Μόλις έρχομαι από άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και ίσως εδώ έχετε προχωρήσει κάπως γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε. Έχω λοιπόν να πω τα εξής. Έχουμε ενώπιον μας μια κατάσταση σημαντικής πίεσης πίεση επί των απασχολουμένων στον τομέα των μεταφορών. Γνωρίζουμε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ανοιχτή αγορά εργασίας στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, εργασίας, της αγωνίας αγοράς μάλλον. Και πολύ καλά κάνουμε. Όμως στη βάση αυτή οφείλουμε να σεβαστούμε την τήρηση των ελάχιστων προτύπων προστασίας των εργαζομένων στο εργατικό δίκαιο. Αυτό αποτελεί μια απόλυτα αναγκαία βάση για να μπορούν ε, να επωφεληθούν όλοι από την ανοιχτή αυτή αγορά. Όταν πρόκειται για δίκαιο της εργασίας, βεβαίως, πρωτίστως οφείλει να λάβει κανείς υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικά εθνικά συστήματα και καμιά φορά υπάρχουν και ανταγωνισμοί όχι μόνο στη βάση των μισθών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων συνθήκων εργασίας στη βάση των εθνικών δικαίων στις διάφορες χώρες μελική. γι' αυτό είναι απολύτως αναγκαίο το υφιστάμενο δίκαιο να τηρεί και να επιτρέπει τον έλεγχο των ελάχιστων αυτών προτύπων. Τα λέω αυτά διότι είναι η δική μας αξίωση. Τώρα, για το ίδιο το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι για τα ε, λόγω των λόγων που εξήγησα μόλι πριν, είναι σημαντικό να ισχύσουν οι κανόνε ήδη από την πρώτη μέρα. Αλλιώς υπονομεύουμε το σύστημα. Πρόκειται για μια απέτηση ώστε να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός επί ε, ίσης Είναι σημαντικό ωστόσο ολόκληρη η Επιτροπή Απασχολήσεως να συμφωνήσει. διότι η οδηγία απόσπαση εργαζομένων θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις μεταφορές. Αν ρωτήσει κανεί τώρα του οδηγού των φορτηγών αυτοκινήτων σχετικά με τι συνθήκε εργασία του, μαθαίνει πράγματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ορομίσιο που φτάνει τα 3,5 ευρώ. Καμιά φορά οι άνθρωποι κάθονται στο τιμόνι 15 ώρες στη σειρά. Περνούν ολόκληρο μήνα όπου ε, διαβιώνουν μέσα στην, ε, στον θάλαμο του φορτηγού αυτοκινήτου. Ορισμένοι από εμά τα είδαν αυτά και στην πράξη. Πρόκειται για συνθήκες οι οποίες δεν είναι αξιοπρεπείς εν τέλει για τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας των μεταφορών είναι από τους πιο ευάλωτους τομείς και επιβαρύνονται οι οδηγοί και μάλιστα ε, εννοώ εδώ τους οδηγούς αμφωτέρων των φίλων, διότι υπάρχουν και πολύ λίγες βέβαια γυναίκες οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων. Εν πάση περιπτώσει, αν αρχίσουμε τώρα να προβλέπουμε εξαιρέσεις θα φτάσουμε να φτιάξουμε ένα ελβετικό τυρί, ολοτρύπες δηλαδή. Ένα σύστημα το οποίο θα οδηγήσει ad absurdum. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε το σύστημα έτσι. Για μένα είναι σημαντικό στα πλαίσια αυτά να τονίσω ότι δεν πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ χωρών με χαμηλό εισόδημα και χωρών με υψηλό εισόδημα. Αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι να είναι δίκαιες οι συνθήκες εργασίας για όλους τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων. Ούτως ή άλλως η αγορά αυτή έχει απελευθερωθεί εντελώς και συνήθως στα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούν άνθρωποι που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Γι' αυτό θα πρέπει να απορρίψουμε το 8 παράγραφος 2, την εξαίρεση δηλαδή, του τομέα των μεταφορών και αντιθέτως να προβλέψουμε αυστηρότερους ελέγχους κατά την εφαρμογή της οδηγίας απόσπασης εργαζομένων. Ευχαριστώ. Thank you. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Μακ Ιντάιερ της Ευρώπης, μάλλον της, συγγνώμη, της ομάδας ECR, μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Μαρτίνα που ε, συνέταξε την, το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Εμείς ε, δουλεύουμε αρκετό καιρό τώρα για την απόσπαση των εργαζομένων και έχουμε εξοικειωθεί πλέον με το θέμα. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα η σαφήνεια της προσέγγισης της εισηγητρίας μας και ε, τη βρίσκω εξαιρετική. Μου αρέσει πολύ επίσης η αιτιολόγηση που προβλέπει η Μαρτίνα ότι οι κανόνες δηλαδή, οι κανόνες εφόσον είναι ασαφείς και δεν εφαρμόζονται επαρκώς δεν οδηγούν σε προστασία των εργαζομένων. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία ε, για όλους τους, ε, για όλους τους φακέλους του τομέα των μεταφορών να εξασφαλίσουμε δηλαδή ε, δίκες συνθήκες, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και βεβαίως και ελευθερία των επαγγελματιών και επιχειρηματιών να προσφέρουν διαμεθοριακές υπηρεσίες. Μέρος της ενιαίας αγοράς που ακόμα δεν έχει πραγματικά ολοκληρωθεί είναι η ενιαία αγορά υπηρεσιών. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικές όταν θεσπίζουμε κανόνες σχετικά για να μην προσφέρουμε τέλει αντικίνητρα στους ε, επιχειρηματίες, στους αυτούς που προσφέρουν υπηρεσίες δηλαδή. Είναι σημαντικό εταιρείε από την Ανατολική Ευρώπη να μπορούν να λειτουργούν και στη Δυτική και βεβαίω και το αντίστροφο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που επιβάλλουμε στις χώρες μέλη. Ταυτόχρονα, επιθυμώ να αποφύγουμε να φτιάξουμε ένα χώρο όπου μπορούν να επιβάλλουν προστατευτικά μέτρα από την πίσω πόρτα οι χώρες μέλη. Πρέπει να είναι σαφές ότι ε, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών από όλους τους ενδιαφερομένους. Υπάρχουν τμήματα της προτάσεως της Επιτροπής που είναι προβληματικά. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής να επιβληθούν έξτρα απαιτήσει στις χώρες μέλη ώστε να περιλάβουν διάφορους, ε, διάφορους ελέγχους συμμόρφωσης ε, roadside checks καθώς ε, δηλαδή οδικούς ελέγχους αλλά και ελέγχους της εγκαταστάσεις κτλ. Είναι ένα τέτοιο παράθυρο. Γι' αυτό και υποστηρίζουν την πρόταση της εισηγητρίας να μειωθούν τα διοικητικά βάρη. Νομίζω επίσης και νομίζω ότι όλες συμφωνήσαμε ότι η ειδικότερη νομοθεσία, ο λέξη σπετσιάλης, έχει σημασία εν προκειμένου και να φροντίσουμε να αποφευθούν οποιασδήποτε περιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τις νέες προτάσεις για την απόσπαση των εργαζομένων, δηλαδή την οδηγία. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ότι το timing, ο χρονισμός των ρυθμίσεων για το τμήμα των μεταφορών θα πρέπει να περιληφθεί στον Lex Specialis. Ξαναλέω για τις μεταφορές. Για να μην υπάρξει κενό νομοθεσίας. Διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ωστόσο, ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι στις μεταφορές καλύπτονται από τις προβλέψεις της ειδική νομοθεσίας, την οποία προωθούμε στη βάση του σχεδίου της Μαρτίνα. Με λίγα λόγια, με εντυπωσιάζει πραγματικά η ποιότητα της εργασίας και την υποστηρίζομαι απολύτως. Thank <coughs> you, Patrick. Ευχαριστούμε. Επόμενο δεν είναι εδώ. Κανείς από την ΚΟΕ. και τότε πράσινη, όχι. Δεν είναι εδώ. Δεν βλέπω κανένα άλλος να παίρνει το λόγο από τους πράσινους. Ρώσα Νταμάτο, από το EFTD. Α, ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως εντόπισε και η συγκήτριά μας, οι ισχύουσες διατάξεις για θέματα απόσπασης δεν επαρκούν για τον υψηλό βαθμό κινητικότητας που διέπει τον κλάδο των οδηγών. Πολλέ φορέ έχουμε να κάνουμε με καταστάσει που δεν επιτρέπουν στου οδηγού να εκτελέσουν σωστά τη καθηκοντά του. Διότι δημιουργούνται διαφορετικά πλαίσια, θέμη του ανταγωνισμού και καταστάσει που δεν μπορούν να ελεγχθούν και να απελευθερωθούν. Η κατάσταση των οδηγών δεν μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση εργαζομένων σε άλλου κλάδου δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κράτος μέλος υποδοχής. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε διαφορετικά την έννοια της απόσπασης. Διότι για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν της διέλευσης και του περάσματο των σύνορων από την πρώτη μέρα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για τη διέλευση θα πρέπει να ορίσουμε ένα χρονικό όριο και να μην γίνει αυτό πρόσχημα για ε, παράνομο καμποτάζ. Ένα επίσης άλλο σημαντικό θέμα είναι να ε, φροντίσουμε για την γρήγορη ταχεία χρήση του εφιού ταχογράφου καθώς και του συστήματος GNS για να διαθέτουμε πληροφορίες για το τι γίνεται καθοδόν, για το εμπόρευμα που έχει στο φορτίο του ενός οδικός, για τον τελικό προορισμό. Όταν τα στοιχεία αυτά είναι ψηφιοποιημένα εξάντε και post, θα μπορούμε να γνωρίζουμε πλήρω τι δράσει έχει κλειώσει ένα οδηγό για μια επιχείρηση. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία, που θα μπορεί να, να ελέγξει τι αμοιβέ των οδηγών και το τι λαμβάνουν οι επιχειρήσει. Αυτό Αυτά είναι μερικά από τα σημεία στα οποία θα συνεισφέρω με τις τοπολογίες μου για να εμπλουτίσω την πρόταση θα θέλαμε να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους στη δουλειά τους και ταυτόχρονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας να τις προστατεύσουμε από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μαρτά και ευχαριστώ τη Μαρτίνα πάνω απ' όλα για τη δουλειά που έχει κάνει που είναι σε βάθος για να εξετάσουμε το θέμα του καμποτάζ. Όμως πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ήδη από το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήξερε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που είναι τα εξή. Οι συνθήκε εργασία των οδηγών, οι ρυθμίσεις και ο θέμητο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μεταφορείς Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Η ευθύνη είναι μεγάλη λοιπόν και όσον αφορά τις αμοιβέ και την κοινωνική προστασία των οδηγών. Σας υπενθυμίζω ότι οι ίδιες ώρες, το ίδιο φορτηγό στους ίδιους δρόμους με το ίδιο εμπόρευμα έχουν διαφορά στην τιμή 8 με 30 ευρώ την ώρα ανάλογα με το αν ο οδηγός ε, είναι από την μία από την άλλη εταιρεία, ανάλογα από πού προέρχεται. 300 με 3.000 ευρώ το μήνα είναι ο καθαρό μισθό ενό οδηγού στην Ευρώπη. Και όταν σταματήσουμε 100 φωτικά διαπιστώνουμε ότι τα 30 κάνουν παραβάσεις. Οπότε πρέπει να το πούμε. Οι ταχογράφοι καταγράφουν 28 μέρες το μήνα. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρχει πάντα ένας εκπρόσωπος εταιρείας στην χώρα υποδοχής για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση και να μην γίνονται απάτε. Φυσικά και θέλουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Οι προθεσμίε πρέπει να μειωθούν. Οι συμπατριώτε μα δεν μπορούν να καταλάβουν πω χρειάζονται τρει μέρε για να πάρει κανεί βασικέ πληροφορίε για ένα φορτηγό και έναν οδηγό που κυκλοφορεί στους δρόμου μα. Ενώ σήμερα μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, σε ένα χάρτη τη διαδρομή, η αστυνομία θέλει τρει μέρε. Μα γίνονται όλα αυτά πολύ εύκολα με τα GPS, οπότε δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια για τους ταχογράφους και την ανταλλαγή δεδομένων. Εμείς θέλουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Τέλος. Το ξέρετε, θέλουμε οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν και να εφαρμόζονται από όλους από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί μια οδηγία για τις οδικές μεταφορές, αλλά μόνο η οδηγία με του, για τους απασπασμένους πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους. Αλλιώς αυτή η διαδικασία δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μεθαύριο για τους λουλουδάδες, αντιμεθαύριο για τους χτίστες και το καθεξής. Εσείς αθνείστε τις τρεις μέρες, κύριε Συγκήτρια, δεν θα εφαρμοστεί και θα εμποδίσει τη δίκηση για τις επιχειρήσεις. Όμω πρέπει να αποφεύγονται καταχρήσεις. Το φορτηγό θα γυρνάει στη χώρα προέλευση του φορτηγού στο τέλος της ε, διαδρομή του. Ο οδηγό θα επιστρέψει επίση σπίτι του. Αλλιώ δεν πρόκειται για διεθνεί μεταφορέ, αλλά για θέμετο ανταγωνισμό. Αντί να έχουμε λοιπόν ένα σταθερό τριών ημερών, πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία του ταχογράφου και του GPS, που μας λέει πού βρίσκεται ανα πάσα στιγμή το φορτηγό και για να αποφύγουμε το αθέμητο καμποτάζ ε, στηρίζουμε να υπάρχει υποχρεωτική εβδομαδία επιστροφή στην χώρα τους και των φορτηγών και των οδηγών τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κύριε Πυρίνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Όχι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Δυστυχώς δεν προβλέπονται τα βουλγαρικά παρά μόνο σήμερα το απόγευμα. Μόνο σήμερα το απόγευμα προβλέπονται τα βουλγαρικά, όχι σήμερα το πρωί. Μα έχουμε και την Προεδρία το απόγευμα, λέει ο κ. Πυρίνσκι. Σήμερα το απόγευμα προβλέπεται, λέει η Πρόεδρος. Συνεχίζει ο κ. και στα αγγλικά. Όσον αφορά τι δραστηριότητε αυτέ λοιπόν που έχουν να κάνουν με την απόσπαση εργαζομένων στι μεταφορέ για τι περισσότερε χώρε μέλη και για τη Βουλγαρία το λέω αυτό, υπάρχουν κανόνε που εφαρμόζονται που είναι διαφορετικοί από του γενικού και αυτό έχει να κάνει τόσο με τι εσωτερικέ όσο και με τι ε, διεθνεί αποσπάσει. Συνεπώς η προσπάθεια, οι γενικοί κανόνες να εφαρμόζονται όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων βάσει της οδηγίας 96 είναι κάτι το οποίο δεν έχει βάση αλλά και δημιουργεί κίνδυνο για χάος στις διεθνείς ε, εμπορικές μεταφορές τις οδικές και δυσκολίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αρχές ελέγχου. Όσον αφορά το πλαίσιο για τις στάνταρτ ε, εμπορικές μεταφορές, ένα φορτηγό μπορεί μέσα σε μία μέρα να περάσει από πολλά και διαφορετικά σύνορα χωρών. Άρα δεν υπάρχει ορθολογικός τρόπος να καθορίσουμε για ποια περίοδο και πώς θα αποδειχθεί ότι συμμορφώνεται ή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας απόσπασης. Βάσει της νομοθεσίας όπου της χώρας όπου βρίσκεται την κάθε χωριστή στιγμή ο οδηγός. Οπότε, Όσον αφορά τις αλλαγές που προτείνει η συγκήτρια, θα αποκλείσουν την εφαρμογή της οδηγίας 96 στις περίπτωσης διακομετα... μυστικών ε, μεταφορών και διεθνών μεταφορών είτε των κάργο είτε των επιβατικών εκτός από την περίπτωση του καμποτάζ όπου θα πρέπει να ισχύει η νομοθεσία της χώρας όπου έχει καταγραφεί, έχει την έδρα της η κάθε εταιρεία. Οι προτάσεις για το καποτάζ λένε να εφαρμόζονται οι κανόνες της οδηγίας απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή όμως η εταιρεία συμμετέχει και στην εσωτερική αγορά της χώρας υποδοχής. Η προσπάθεια τώρα να υπάρξουν διάφορες εξαιρέσεις όπως προτείνεται, μάλλον θα δημιουργήσουν δυσκολίες και διαφορετικές ερμηνείες και εφαρμογή των κανόνων. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα για την βελτίωση των ελέγχων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι, οι προτάσεις της Επιτροπής δικαιολογούνται απόλυτα. Δεδομένου των δυνατοτήτων που υπάρχουν και οι περιπτώσεις ε, να χρησιμοποιηθεί στραβά ο ταχογράφος και να δείξει στραβά αποτελέσματα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τους ευφύς ταχογράφους, τους οποίους δεν θα μπορεί κανείς να τροποποίηση καταβούληση. Η προσπάθεια επίσης να υπάρξει επιπλέον νομοθετική ρύθμιση και που λέει ότι τα έγγραφα θα τα κρατάει ο οδηγός και θα μπορεί να τα δώσει σε περίπτωση ελέγχου και θα έχει και αντίγραφα των συμβολέων του ε, αποδείξει για τις πληρωμές του και κτλ. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκω ότι είναι εντελώ δυσανάλογα. Θα πρέπει η εταιρεία να ελέγχεται και όχι ο οδηγός. Οι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανάλογα με το που έχει την έδρα της επιχείρηση κάθε φορά. Συνεπώς, οι προτάσεις της εισηγητρίας είναι ένας καλός συμβιβασμός. Εφόσον τα έγγραφα αυτά θα δίνονται άπαξ και ζητηθούν, Και θα πρέπει να τα δίνουν οι εκπρόσωποι της εκάστοτε επιχείρησης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Κατόπιν όλων αυτών, προτείνω να στηρίξουμε καταρχήν την προσέγγιση της εισηγήτριας στον λόγο θέμα και τις αντίστοιχες τροπολογίες και θα υποβάλω και εγώ τροπολογία. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, με συγχωρείτε που δεν έχουμε βουλγαρικά. Έκανα μόνος μου την μετάφραση. Ναι, την κάνατε τέλεια τη μετάφραση. Και τώρα λόγο στην κυρία Λόπε Φοντανιέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω να κάνω δύο σχόλια όσον αφορά την απόσπαση, μια που είμαι και εγώ η συγγήτρια για ένα αντίστοιχο θέμα. Θέλω να μιλήσω για τις επιπτώσεις της οδηγίας πάνω στους οδηγούς. Το περιθώριο αυτό των τριών ημερών σε ένα μήνα δεν φτάνει, γιατί δεν προσφέρει αρκετό χρόνο στον οδηγό για να επιστρέψει στη χώρα του, κυρίως την περίπτωση που πρόκειται για περιφερειακές χώρες. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πλήττονται κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το διακομιτιστικό εμπόριο πρέπει να εξαιρείται, συμφωνώ, και επανέρχομαι στο θέμα των ημερών, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών, 5-7, που να είναι διαδοχικές. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι απαιτήσει πρέπει να καλύπτουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους οδηγούς εφόσον ξεπεραστεί αυτό το διάστημα γιατί δεν είναι το ίδιο να χρησιμοποιεί έναν οδηγό ένα χρόνο μια επιχείρηση ή άλλο χρονικό διάστημα. Οπότε πρέπει να λυθει και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό για μένα να, αποτιμήσω, να, να αποτίσω φόρο τιμής στην εργασία της ε, εισηγητρίας. Και για μας είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφέστερα οι κανόνες, ώστε αφενός να έχουν τη δυνατότητα και οι επιθεωρητές, ελεγκτές, να κάνουν τη δουλειά τους και επομένως να κάνουν σωστά τους ελέγχους. Πράγματι έχει ιδιαιτερότητες στο τομέα των μεταφορών και είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Διεθνείς μεταφορές, καμποτάζ, εθνικές αγορές, ορισμένες επιχειρήσεις άλλωστε ειδικεύονται στην ανάμιξη των διαφόρων μεταφορών ώστε οι έλεγχοι τελικώς δυσχεραίνονται σημαντικά Όλοι, μάλλον όλες οι τροπολογίες που ε, θα καταστήσουν τους ελέγχους αποτελεσματικότερους θα με βρουν σύμφωνο και στην Επιτροπή Μεταφορών όπου επίσης συμμετέχω ως μέλος. Τώρα βέβαια για τις εξαιρέσει που θα αρχίσουν και που θα τελειώνουν. Εάν εξαιρέσει κανείς ένα τομέα, ας πούμε το transit, τη διαμετακόμιση. Βέβαια, για τη χώρα μου, το Λουξεμβούργο, κοιτάξτε, διασχίζουν ε, τα φορτικά του Λουξεμβούργο μέσα σε λιγότερο από μια ώρα. Για πολλές όμως μεγάλες χώρες και το transit είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, εάν εξαιρεθεί δηλαδή από την οδηγία. Πρέπει λοιπόν να ρίξουμε το βάρος μας στην αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού. Και αυτό το πρέπει να αποτρέψουμε για την εξαίρεση ή αφαίρεση τέλος πάντων από τη γενική οδηγία σκεφτείτε ότι ενδέχεται να φτιάξουμε ένα κενό Προτιμώ λοιπόν να παραμείνουν οι οδικές μεταφορές στη γενική, στα πλαίσια της γενικής οδηγίας, οι ιδιαιτερότητες δε του τομέως να ρυθμιστούν μέσω του Lex Specialis. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μωράν Σαρτιέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που ασχολούμαστε με το θέμα των ε, αποσπασμένων εργαζομένων για οποιοδήποτε κλάδο και αν πρόκειται. Ευχαριστώ την κυρία Τζαμπάλοβα για τη δουλειά της. Πρόκειται για δουλειά εξαιρετικά δυσχερή για να προσαρμόσουμε την οδηγία περί απόσπασης σε λέξ σπεσιάλης για τον τομέα των μεταφορών. Ε, συμφωνώ σε πολλά με την κυρία Τσαμπάλοβα και με τις προτάσεις της, ιδίως ως προς τη σημασία εφαρμογής των όσων ισχύουν ε, για την απόσπαση σε σχέση με το καμποτάζ. Το καμποτάζ είναι πραγματική μορφή ανταγωνισμού για τις τοπικές επιχειρήσεις και πρέπει στην εσωτερική αγορά οι επιχειρήσεις να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες ως προς τις αμοιβέ και οι μισθωτοί να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Αυτό είναι βάση για τον ε, σεβασμό, την τήρηση μιας αρχής που αποφασίστηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιούνκερ για ίση δουλειά, ίση αμοιβή. Ε, επίσης, συμφωνώ ότι η απόσπαση δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις δράσεις διέλευσης, ε, εφόσον δεν υπάρχει εμπορική δραστηριοποίηση σε επικράτεια τους μέλους. Δεν πρόκειται για άμεσο ανταγωνισμό. Όμως, αυτό δεν ισχύει πάντοτε, όπως γνωρίζουμε, και κάποιες δράσεις είναι λίγο υπόγειες, λίγο ανάμεικτες, οπότε εκεί γίνεται δύσκολο να κάνει κανείς τον έλεγχο και περνάμε σε ζώνες λίγο πιο θολές. Ε, κατά τα άλλα, ό,τι αφορά τη διεθνή κυκλοφορία, δεν θα συμμεριστώ την ε, οπτική γωνία της εισηγητρίας, που κατά τα άλλα τη σέβομαι βεβαίως, η οποία θέλει να εξαιρεθούν αυτέ οι δραστηριότητε από το σύστημα περί απόσπαση. Εάν υπάρχουν εμπορικέ δραστηριότητε σε μια χώρα, θα πρέπει οι κανόνε να είναι ίδιοι για τι εταιρείε και τι επιχειρήσει. και τα δικαιώματα τα ίδια για του εργαζομένου. Αυτό είναι ο στόχο τη αναθεώρησης τη οδηγία περί απόσπαση. Και θα έπρεπε να είναι και στόχο τη Lex specialis, του ειδικού νόμου, ε, ακόμα και αν υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, καταστάσεις. Αυτή η ισότητα των δικαιωμάτων επιτρέπει και η ισότητα μεταχείριση. Αυτό είναι και η βάση, ε, τα θεμέλια που θέλουμε να δημιουργήσουμε για την κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν το καθεστώ ε, τη απόσπαση να ισχύει και για τι διεθνεί μεταφορέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει προθεσμία τριημέρου μέχρι να ε, εφαρμοστεί το σύστημα περί απόσπαση. Μπορούμε να χαιρετήσουμε την προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να βρει μια συμβαστική λύση, αλλά η εφαρμογή αυτού του μέτρου φαίνεται να είναι δύσκολη. Θα ήταν πολύ απλούστερο το σύστημα της απόσπασης να ισχύει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα. Οι υπόλοιπε προσπάθειε αιτιολόγηση και εξήγηση είναι άνευ λογοκαιτία, διότι όλοι ξέρουν σε αυτή την αίθουσα, όλοι, ότι ε, ο ταχογράφο ενημερώνει αμέσω. Και μπορεί κανεί να έχει αυτομάτω όλε τι απαραίτητε πληροφορίε, χάρη στον ταχογράφο, ε, μέσω των ελέγχων για το σύνολο των ε, φορτηγών των βαρέων οχημάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος αναβολής. Δεν χρειάζεται η αναπομπή στις ελληνικές καλένδες αυτού του ε, θέματος, εφόσον έχουμε τεχνολογικά μέσα που το επιτρέπουν αυτομάτως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή των κανόνων, μπορούμε να παραμείνουμε σε ένα θολό τοπίο από νομικής πλευράς ε, καθώς δεν υπάρχει ειδικό νόμος, lex specialis, και σας θυμίζω ότι για την οδηγία της απόσπασης ζητάμε εδώ και 22 μήνες, πρόεδρε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ε, η lex specialis έχει αρχίσει ήδη να μελετάτε. Τι θα γίνει, θα την ολοκληρώσουμε την νομοθεσία αυτή πριν τις ευρωεκλογές το 2019. Ποιος εδώ μπορεί να το διασφαλίσει. Κανείς και καμία. Πρέπει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο περατωμένο κείμενο. Ίσως τα καταφέρουμε, αλλά ίσως και όχι. Τι θα γίνει λοιπόν εάν ε, ο ειδικό νόμος δεν αρχίσει να εφαρμόζεται πριν τις ε, εκλογές του 2019. Πώς θα έχει διαμορφωθεί το σώμα μας μετά το 2019. Πότε θα το περατώσουμε. Πρέπει να σας πω πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά τη θέση μου περί του θέματος, ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ορθολογιστές εφόσον θέλουμε λέξη σπεσιάλης, πρέπει να ψηφιστεί εδώ και η αναθεωρημένη οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων να εφαρμοστεί στον τομέα των οδικών μεταφορών. Όχι όμως η οδηγία του 96, από μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 15 κράτη-μέλη με μισθούς και διαφορές που πήγαιναν από το 1 στο 3 όχι για σήμερα, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτό το πεδίο. Ναι, λέξ specialis, η κατάσταση να είναι όμως πια καθαρή και να επιτρέπεται να γίνουν σωστά οι έλεγχοι και οι παληθεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ο κύριος Καλβέ Τσαμπόν είναι ο επόμενος, αλλά δεν είναι εδώ. Η κυρία Σόιντροβα είναι και θα την ακούσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να τοποθετηθώ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Προσωπικώς υποστηρίζω τις ε, προτάσεις της εισηγήτριας. Και έχω και δικές μου προτάσεις να κάνω. Θα τις υποβάλλω μέσω των τροπολογιών. Το πρώτο τμήμα αφορά την αλλαγή για τους κανόνες απόσπασης των εργαζομένων γενικώ και ειδικώ στον τομέα των μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει σε έλεγχο των κοινωνικών προποθέσεων που ισχύουν για τους εργαζομένους αυτούς και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να τα παρακολουθήσει αυτά. Δεν ακούω κανένα να λέει ότι χρειαζόμαστε διασυνοριακά επαγγελματικότερου ελέγχου. Η πρότασή μου θα φροντίσει να το καλύψει αυτό. Δεύτερο τμήμα για του τομεακούς κανόνες. Εκεί έχω απογοητευτεί κάπω, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ξεκάθαρα και το είπαμε και εμείς κατά τη συζήτηση περί απόσπασης ότι χρειαζόμαστε lex specialis. Χρειαζόμαστε νομοθεσία ειδική στοχευμένη για τον τομέα των μεταφορών. Η πρόταση εδώ περιορίζεται αρκετά με την προθεσμία των τριών ημερών. Δεν πρέπει να παραμείνουμε τόσο προσιλωμένοι σε αυτή την προθεσμία του τριημέρου. Πρέπει να σκεφτούμε πώς υπολογίζουμε το χρόνο και τι σημαίνει αυτό γενικότερα για αυτόν τον κλάδο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είμαι υπέρ της επιμήκυνσης της παράτασης αυτής της περίοδου για να μπορούμε να έχουμε ικανοποιητικέ διεθνεί μεταφορέ. Υπό αυτήν την έννοια θα υποβάλω και τι δικέ μου τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Μπαλά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλό είναι να μην συγχαίουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Η δουλειά ενός οδηγού στους αυτοκινητοδρόμους είναι διπλή η μεταφορά από τη μία, οι εμπορικές δράσεις από την άλλη, φόρτωση, μεταφόρτωση και το καθεξής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στο πρώτο επίπεδο, νομίζω ότι η κυρία Δεμπάλοβα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ιδίω ό,τι αφορά το καμποτάζ. Ναι, για το θέμα του καμποτάζ νομίζω ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εμπορικέ δράσει, οπότε πρέπει να υπάρχει σαφή νομοθεσία. Ε, για και να ισχύουν όσοι ισχύουν για την απόσπαση των εργαζομένων. Διότι αυτοί οι κανόνε επιτρέπουν ακριβώ αναρμόνιση των κοινωνικών προτύπων και αποφεύγουν το κοινωνικό ντάμπινγκ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι διαθέσει μεταφορέ, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το τι ανήκει σε μεταφορέ ακριβώ, ε, όταν ο οδηγό οδηγεί απλώ δηλαδή το όχημα και τι είναι εμπορική δράση. Εδώ νομίζω ότι πράγματι πρέπει να κάνουμε τη σωστή διάκριση. Όταν ένα οδηγό απλώ διασχίζει μια χώρα, ε, δεν έχει πολύ νόημα για λίγε ώρε να ισχύουν οι κοινωνικοί κανόνε του κράτου αυτού. Όμω, εάν εκεί αυτό ο οδηγό έχει μαζί του κάποιον άλλον εργαζόμενο, ο οποίο θα κάνει την εκφόρτωση και τη μεταφόρτωση, εκεί θα πρέπει να ισχύουν οι κοινωνικοί κανόνε τη χώρα και να ισχύουν ε, τα κοινωνικά πρότυπα. Η οδηγία λοιπόν περί απόσπαση θα μπορούσε αυτό να το καλύπτει και γνωρίζουμε ότι. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ απλά όλο αυτό. Έχουμε τον ταχογράφο. Ε, υπόθηκε επανειλημμένο τεχνικώ έχουμε τα μέσα. Δεν λείπει λοιπόν πλέον κάτι πέρα από την πολιτική βούληση στην ε, χώρα μας. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει τις νέες γενιές να περιμένουν τόσο πολύ ε, για να δουν το αποτέλεσμα που, δεν, ε, που κινδυνεύουμε να μην πετύχουμε. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να φτάσουμε σε κάτι ικανοποιητικό και για τους κανόνες της απόσπασης. Και κάτι ακόμη, οι προθεσμίες, το είπε και η συγκήτρια, Η συγγήτρια για το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων, κυρία Μωράν Σαρχέ, έχει δίκιο. Πρέπει να καλύψουμε το νομικό κενό. Εάν δεν υπάρχει λέξη specialis, θα πρέπει οι οδηγοί παρόλα αυτά να καλύπτονται και θα πρέπει να ισχύσει η νέα νομοθεσία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ιδάλω υπάρχει στράβλωση από τη μια μεταξύ όλων των εργαζομένων και των κανόνων που του διέπουν και από την άλλη των οδηγών. Νομίζω ότι μάλιστα θα μπορούσε κανεί και να προσφύγει σε αυτή την περίπτωση, αν γίνει κάτι τέτοιο. Και κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι λίγο από αυτό που είπε ο συνάδελφος από το Εθνικό Μέτωπο προηγουμένω, από το Front National. Γιατί αγωνιστήκατε κατά όλων των νομοθεσιών που τείνουν να εναρμονίσουν τους κοινωνικού κανόνες για τους εργαζόμενους, θεωρώντας ότι δεν έχει δουλειά εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει μόνο τα εθνικά κράτη να το κάνουν. Τι σέβομαι τη θέση σα, δεν ταυτίζεται με τη δική μου, αλλά το καταλαβαίνω. Σήμερα ε, σφετερίζεστε τα επιχειρήματα της ε, νομοθεσίας για την απόσπαση των εργαζομένων που σας φαίνονται αξιοθαύμαστα ε, από αυτή την σκοπιά και ξαφνικά μας λέτε ότι δεν πήγε αρκετά μακριά η δουλειά της συγκέντρωση ε, της κυρία Τζαμπάλοβα. Εδώ υπάρχει μια σαφής αντίφαση και ένα παράδοξο που κάποτε μπορεί να λυθεί. Ευχαριστούμε. Ο κατάλογος μου λέει να περάσουμε ευθύ αμέσως στο επόμενο σημείο. Η είναι ο κύριος Μπαχ. Ξέχασα κάποιον. Α, με συγχωρείτε βεβαίως κυρία Τζαμπάλοβα. Ε, βέβαια πρέπει να δευτερολογήσετε. Γιατί και στο επόμενο σημείο τη ημερήσια θα ξαναζητήσετε το λόγο. Ναι, ναι, απλώ λιγάκι να αντιδράσω και να έχω την ευκαιρία να τα συνοψίσω λίγο. Να ευχαριστήσω όλου για τι συνεισφορέ του, διότι νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε διαφορετικέ σκοπιέ και βεβαίω θα τα λάβω όλα υπόψη ε, τη στιγμή τη επεξεργασία των συμβιβαστικών. Ανυπομονώ λοιπόν να δω τι συμβιβαστικέ λύσει ε, και το τι θα προκύψει και τι συζητήσει με του σκιώδε. Υπάρχουν πολλέ δηλώσει με τι οποίε διαφωνώ. Δεν θα πω τώρα με ποιον ακριβώ ε, διαφωνώ και ποιον συμφωνώ. Απλώ να σα θυμίσω ένα-δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κυρία Ρέγνερ, να σα θυμίσω ότι ψηφίσαμε στην Επιτροπή μα για την απόσπαση των εργαζομένων και την οδηγία αυτή τα θέματα μεταφορών να παραπενθούν σε λέξ πεσιάλη. Το ψηφίσαμε όλοι. Ήταν αποτέλεσμα τη ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ε, το τι θα γίνει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο θα δούμε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν το θέλουμε στην Επιτροπή μα γιατί ψηφίστηκε. Δεύτερον, πρέπει να δούμε το εργαλείο αυτό από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Γι' αυτό πρότεινα αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση, διότι είναι πολύ σαφέ και απλό, εύληπτο και το κοιτάζει το θέμα από διαφορετικέ ε, προοπτικέ, από διαφορετικέ σκοπιέ. Ποιο είναι το πρόβλημα, Όλοι το είπατε με τον τον άλλο τρόπο. Ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Θέλουμε να α, αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Συμφωνούμε όλοι. Θέλουμε να αποφύγουμε τι καταχρήσει. Θέλουμε να αποφύγουμε τον διοικητικό φόρτο για τι εταιρείε. Το γραφειοκρατικό, το γραφειοκρατικό δηλαδή. Θέλουμε να αποφύγουμε όλου αυτού του παράγοντε που προκαλούν τον αθέμητο ανταγωνισμό οι οδηγοί να καλυφθούν καλύτερα από την γνωμοδότηση του κυρίου Μπάχα, τα ακούσουμε τώρα. Αλλά να τι προκαλεί αθέμη τον ανταγωνισμό. Ο, το καμποτάζ σε κάποιε περιπτώσει. όλοι το αναφέρατε. Νομίζω όλοι συμφωνούμε, όλοι συμφωνούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Απλώ να σα πω ότι η συλλογιστική τη εκθεσή είναι λίγο διαφορετική. Ήθελα να απομακρυνθώ από αυτή την καταμέτρηση ημερών, διότι να ξεκινήσει κανεί και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαστε όλοι φοβερά ε, πείσμονε. Εάν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για τον αριθμό των ημερών, ο ένα θα θέλει τρει, ο άλλο πέντε, ο άλλο είκοσι και ο άλλο όσο να είναι. Δεν θα ξεφύγουμε ποτέ. Η λογική μου λοιπόν ήταν να δούμε τα πραγματικά προβλήματα να ορίσουμε τις διεθνείς μεταφορές ε, με σαφήνεια και να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των εργαζομένων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Ας δούμε τις διαφορετικές προοπτικές. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες, εάν θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε διοικητικό άχθο για τις εταιρείε, ε, πού είναι ο κοινός νου στην εφαρμογή. Δεν θα ξεφύγουμε ποτέ. Θα είμαστε εδώ σε ένα χρόνο να τα συζητάμε και πάλι σε δύο χρόνια θα ξαναβρεθούμε να τα συζητάμε. Δεν έχει λοιπόν όλο αυτό να κάνει με τον αριθμό των ημερών. Δεν έχει να κάνει με το αν κάποιο θέλει τρει μέρε ή είκοσι. Έχει να κάνει με το τι θέλουμε να κάνουμε για την ενιαία αγορά. Και το τελευταίο μου σχόλιο, και σε ευχαριστώ Ελιζαμπέτ που το ανέφερε, η θέση σε ισχύ. Είναι πραγματική πρόκληση. Το ανέφερα στην αρχή της, ε, στην πρώτη μου παρέμβαση. Θα ήθελα όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτά τα διαφορετικά θέματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώ θα φροντίσουμε την θέση σε ισχύ και για την αναθεώρηση τη οδηγία περί απόσπαση εργαζομένων και για την Lex Specialis. Ναι, Πρόεδρε, θα ξαναμιλήσω, διότι είμαι συγκίτρια και στα επόμενα δύο θέματα. Βρίσκω ότι αυτή η φάκελη είναι αλληλένδετη και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς διασυνδέονται και ποια είναι η κοινή λογική που τους διέπει. Ευχαριστούμε. Το χρονοδιάγραμμα είναι συνδεδεμένο βέβαια για αυτά που εξετάζουμε. Προθεσμία για τροπολογίες για την έκθεση αυτή είναι 30 Ιανουαρίου. «27 και 28 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και μετά θα πάμε στις 15 Μαΐου στην Επιτροπή Μεταφορών. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα ακριβώς έχουμε και για το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και περνάμε ευθύ αμέσω στο επόμενο, γιατί ακριβώς είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζορς Μπαχ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μπαχ. Διαπιστώνω εξ αρχής ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει και θετικά σημεία. Για παράδειγμα, βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις διοικητικές αρχές, βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών. Σημαντική είναι επίσης η διευκρίνηση ότι η εβδομαδιαία ανάπαυση 45 ωρών δεν μπορεί να γίνεται μέσα στον θάλαμο του φορτηγού αυτοκινήτου. Αυτά τα έχει δεχτεί σε απόφασή του και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ίδιο η ιδέα ότι ο οδηγό θα πρέπει να μπορεί να επανέρχεται στην αιστεία του είναι σωστή. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Γι' αυτό εγώ προτείνω ορισμό της αιστεία στα αγγλικά home, το σπιτικό δηλαδή, που να, έχει, να λαμβάνει υπόψη του και τον τόπο διαμονή του οδηγού αλλά και την έδρα της επιχειρήσεω. Από την αρχή θεώρησα ότι οι κανόνες που ισχύουν σχετικά με την ώρα αναπαύσεως ή μάλλον με, την περίοδο αναπαύσεως είναι επαρκής εάν εφαρμόζονται σωστά. Και γι' αυτό στη γνωμοδότησή μου προτείνω να διατηρηθούν οι περίοδοι αναπαύσεως που ισχύουν τώρα. Προσπάθησα επίσης να περιλάβω όλα τα θετικά σημεία μαζί σε ένα τμήμα της εκθέσεως με τον στόχο να βελτιωθεί η εργασία των οδηγών και επομένως και η ασφάλεια των μεταφορών. Φορτηγά αυτοκίνητα κάτω των 3,5 τόνων θα πρέπει επίσης να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα όμως θα πρέπει να εντάσσονται στις ε, προβλέψεις της οδηγίας εφόσον κινούνται σε μια ακτίνα πέραν των 100 χιλιόμετρων από την έδρα της επιχειρήσεως για να μην υπάρχουν στροπλώσεις του ανταγωνισμού. Επίσης, η αποζημίωση για μειωμένες περιόδους αναπαύσεως θα πρέπει να συνδυάζεται και με την εγγύηση της 45ωρης ε, περίοδου αναπαύσεως. Αυτό σημαίνει ότι το αργότερο μετά από 5 εβδομάδες θα πρέπει να υπάρχει περίοδος αναπαύσεως τουλάχιστον 66 ωρών. είτε στο σπίτι του οδηγού είτε σε άλλο τόπο τον οποίο επιλέγει ο ίδιος ο οδηγός. Τροπολογία υπαρθμονετικά. Είναι ρεαλιστικό να απαιτήσει κανείς από τις επιχειρήσεις να οργανώσουν την εργασία τους με τέτοιο τρόπο ώστε οι οδηγοί το αργότερο κάθε πέντε εβδομάδες, ένα μήνα και μια εβδομάδα δηλαδή, να μπορούν να επανέρχονται στο σπίτι τους. Από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι και η ημερομηνία από την οποία και μετά θα εξοπλίζεται το κάθε φορτηγό αυτοκίνητο με τον λεγόμενο F.E. ταχογράφο. Αυτό έχει τονιστεί ήδη πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει το όργανο αυτό. Μιλούμε για πραγματική τεχνολογική επανάσταση. Η ψηφιοποίηση δηλαδή θα πρέπει να εισχωρήσει και στα φορτηγά αυτοκίνητα. Και βλέπω ότι ε, μεγάλες δυσκολίες προκύπτουν σε ό,τι αφορά την ε, τον εξοπλισμό με ε, τους εφείς ταχογράφους. Ε, ο Ιούνιος του 2019 που προβλέπεται για μένα πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε στην νομοθεσία. Αν και προβλέπεται μεταβατική περίοδος 15 ετών. Εγώ προτείνω να μειωθεί αυτή στα 5 έτη. Αυτό να συνδυαστεί και με την μείωση του διοικητικού άχθους των επιχειρήσεων και βεβαίω θα διευκολυνθεί τότε και η εργασία των επιχειρήσεων και των οδηγών. Άλλο θέμα που ήταν σημαντικό για μένα ήταν η ενίσχυση του άρθρου που λέει ότι η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να πληρώνει ούτε καν να πρημοδοτεί στην βάση της διανυόμενης αποστάσεως και του μεταφερόμενου φορτίου. Μέχρι τώρα αυτό ισχύει μόνο εφόσον μια μεταφορά αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Όμως δεν ελέγχονται τα πράγματα αυτά ή δεν είναι και δυνατόν να ελεγχθούν, ώστε οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα να πληρώνουν τους οδηγούς έτσι. Θα συνεργαστώ βεβαίως με τους και ελπίζω να διαμορφωθεί καλά αυτή η συνεργασία. Για μένα είναι σημαντικό να δώσουμε ένα καθαρό μήνυμα. Νομίζω ότι με κοινή προσπάθεια μπορούμε να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στου εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις και για τις αρχές ελέγχου, αλλά βεβαίω και ιδίω για την ε, οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Μπαχ. Τώρα θα προχωρήσουμε να ακούσουμε τους σκιώδει εισηγητέ. Ο κύριος Σούλες Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε στα αγγλικά. Πρώτη γενική παρατήρηση. Εάν δεν μπορέσουμε να επιφέρουμε βελτιώσεις για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τον τομέα των μεταφορών ελκυστικό, έτσι ώστε να προσελκύσει ε, προς τον τούχους οδηγού στο μέλλον. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Μπαχ, εισηγητή, που θεωρώ ότι τα έχει πάει πολύ καλά έως τώρα ε, στην έκθεσή του. Συμφωνώ δε με τι περισσότερε από τι τροπολογίε που έχει καταθέσει ο ίδιο ο κ. Μπαχ. Για άλλα θέματα θα προτείνω και εγώ ορισμένε τροπολογίε, που ωστόσο θα έχουν ε, το ίδιο πνεύμα. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα πράγματα που εγώ θέλω να προχωρήσω περισσότερο από τον ίδιο τον κύριο Μπαχ. Δύο από αυτά θα σα αναφέρω ω παράδειγμα. Θα ήθελα πρώτα ο ευφύης ταχογράφο ε, να εισαχθεί το δυνατόν συντομότερο. Ο ευφύ ταχογράφο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιβολή των ελέγχων και δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην μπορεί να ε, εισαχθεί ήδη από το 2021, να αρχίσει να χρησιμοποιείται σε όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα. Επίσης, ο εργοδότης θα πρέπει να αποζημιώνει τον οδηγό για την επιστροφή στην αιστεία του, ώστε να μην μένει ο άνθρωπος κάπου σε κάποια ξένη χώρα. Χρειαζόμαστε ε, συμβασμού για το φάκελο αυτό που να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των οδηγών σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεργαστώ βεβαίως και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζλοτόφσκι των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εκ μέρους μου ευχαριστίες προς τον κύριο Μπαχ για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Συμφωνούμε όλοι ότι ο επαγγελματίας οδηγός κάνει μια δύσκολη δουλειά και όλοι επιθυμούμε να δούμε οι άνθρωποι αυτοί να αναπάγονται επαρκώς διότι μόνο έτσι θα μπορούν να οδηγούν και με ασφάλεια. Ας μην λησμονούμε ωστόσο ότι ο τομέας αυτός είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητος στις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που εν τέλει οδηγούν σε υψηλότερο κόστος και σε περιορισμούς χρόνου. Ο ίδιος ο κύριος Μπαχ τόνισε ότι δεν υπάρχουν και αρκετοί ε, χωριστάθμευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με μια Γερμανική Ένωση Επαγγελματιών Διαχειριστών Χώρων Στάθμευσης, λείπουν στη Γερμανία, φανταστείτε, 31.000 θέση Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν να περάσουν πολλέ δεκαετίε ώστε να υπάρξουν επαρκείς χώροι στάθμισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε δεκαετίε ολόκληρε μέχρι ότου ε, να ε, φτιαχτούν αυτά. Η δυνατότητα εβδομαδιαία αναπαύσεως μέσα στον θάλαμο του φορτηγού αυτοκινήτου είναι λοιπόν αναγκαία και πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για αυτούς που καλύπτουν μακρές αποστάσεις, το οποίο εν τέλει και αυτό είναι αναγκαίο λόγω της ενιαίας αγοράς. Δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή ο άνθρωπος να αναπαύεται μέσα στον θάλαμο του φορτηγού, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα. Το άλλο θα πρέπει να είναι η maximum περίοδος ε, οδήγησης και η δυνατότητα επιστροφής στην αιστεία του ώστε να μπορεί να αναπαύεται την εβδομάδα παραπάνω από 45 ώρες. Ε, ο εισηγητής ε, έχει τροποποιήσει σημαντικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής, Οδηγίας, της ευρωπαϊκή Επιτροπής συγγνώμη, που προβλέπει κιόλας ότι θα πρέπει να επιστρέφει ο οδηγό στην αιστεία του ανά τρει εβδομάδε. Αυτό όμω δυσχεραίνει πολύ τον προγραμματισμό ίσως χρειάζονται έξι διαδοχικές εβδομάδες ως καλύτερη λύση και να μπορεί να επιλέγει ελεύθερα ο οδηγός που θα περάσει την περίοδο ανάπαυσής του. Τώρα ένα άλλο θέμα είναι η εφαρμοσιμότητα των κανόνων και για τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα κάτω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους που χρησιμοποιούν κυρίως μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να σημάνει ωστόσο σημαντική γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις ε, ΜΜΕ και να αυξήσει το κόστος λειτουργίας τους και μάλιστα δυσανάλογα ανάλογα με, δυσανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Άλλο θέμα είναι η συντομία της ε, περίοδου αναπαύσεως. Τώρα, ε, υπάρχει και το θέμα των εφιών ταχογράφων. Ο συμβασμό που έχει ε, επιτευχθεί με τη σχέδια είναι σημαντικό να διατηρηθεί. Οι ευθύς ταχογράφοι, όπως λένε οι ειδικοί, δεν πρόκειται να λύσουν όλα τα προβλήματα. Το δε κόστο τη εγκατάστασή του στα φορτηγά αυτοκίνητα είναι υψηλό και αποτελεί πρόκληση ιδίω για τι μικρέ επιχειρήσει μεταφόρων. Η προσπάθεια λοιπόν να αλλάξει η πρόταση της Κομισιόν προς την κατεύθυνση αυτή δεν είναι δικαιολογημένη. Υποστηρίζω τον κύριο Μπαχ όταν λέει ότι το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί για να γίνει ασφαλέστερος ο τομέας αλλά και πιο ελκυστικός είναι βασικά το ζήτημα της έλλειψης χώρων σταθμεύσεως και οικονομικής, οικονομικών καταλημάτων, δηλαδή ευθυνών καταλημάτων. Αν αλλάξουν σημαντικά οι κανόνες στην αρχή της διαδικασίας, αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι μεγάλη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και ιδίως από τις χώρες της περιφέρειας. Το δε κόστος θα το αναλάβουν τελικώς οι επιχειρήσεις και το κόστος αυτό θα μεταφερθεί εν τέλει, θα μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες και είμαι πεπισμένος ότι παρά τις διαφορές ε, των θέσεών μας θα καταλήξουμε σε συμβασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε. Μια στιγμή. Ε, yes, it's uh, Η Ματίνα. Ναι, πάλι εγώ. Όλο για σένα μιλάμε εδώ. Η σειρά σου. Είναι καλό γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο θέματα, οπότε είναι καλό που τα συζητάμε έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπαχ για το σχέδιο γνωμοδότησής του, όπως είπα και πριν. Είναι η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο σημείο να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, χρόνο και τα λοιπά. Πάντως, ο τελικός μας στόχος πρέπει να είναι κανόνες που να είναι εφαρμόσιμοι και να μπορούν να δουλέψουν στην πράξη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να αποφασίσουμε κανόνες που να λειτουργούν. Κύριε Μπαχ, χαίρομαι που αναφερθήκατε στην ανησυχία αυτή για τον ύπνο των οδηγών στα φορτηγά του πολύ σωστά λέτε στη γνωμοδότησή σας ότι δεν έχουμε κατάλληλες υποδομές. Οπότε όσο δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές, δεν είναι ρεαλιστικό να απαγορεύσουμε τον ύπνο μέσα στα φορτηγά. Μπορούμε να συστήσουμε τη δυνατότητα να κοιμούνται οι οδηγοί εκτός του φορτηγού, ναι, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια διαθεσιμότητα αλλά πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε υποδομέ. Οπότε πρέπει να είναι μόνο μια σύσταση, κατά τη γνώμη μου, και τίποτα παραπάνω. Χαίρομαι επίση που βλέπω και αλλαγέ όσον αφορά την επιστροφή για την εβδομαδία ανάπαυση στην χώρα τους. Στην πρόταση της επιτροπή μου φαίνεται πολύ αυστηρό. Πρέπει να μπορεί ο οδηγό να επιστρέφει στο χώρο που ο ίδιος επιλέγει δεν πρέπει να είναι οικονομική υποχρέωση για την εταιρεία να πληρώσει κάποιες διακοπές που μπορεί να επιλέξει να κάνει ο οδηγός, αλλά πρέπει να μπορεί να επιστρέψει όπου θέλει και να πληρωθεί για τα έξοδα επιστροφής του στη χώρα του, που θα είναι η μόνιμη διαμονή του οδηγού ή η έδρα της επιχείρησης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό. Δεν είμαι τώρα πολύ πεπισμένη για τα εμπορικά οχήματα, ελαφρά εμπορικά οχήματα αυτά που λέτε, αλλά με τους σκιώδεις εισηγητές να το συζητήσω μαζί σας αν θέλετε. Τέλος, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ελαστικότητα και περισσότερο ρεαλιστικούς χρόνους όσον αφορά την οδήγηση και την αναπαύση των οδηγών. Η περίοδος αναφοράς τεσσάρων εβδομάδων μου φαίνεται εντάξει και για να έχουμε περισσότερη σαφήνεια Νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την επιστροφή του οδηγού στη βάση του, γιατί νομίζω ότι προτείνει τρει εβδομάδε περίοδο αναφορά γι' αυτό η Επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και εκεί να είναι τέσσερι εβδομάδε. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συντονιστούμε πολύ καλά. Πρόεδρο. ευχαριστούμε. Κυρία ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για το έργο του. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά που λέει ο κυρίος Μπαχ. Παρόλο που υπάρχουν κάποια θέματα που θα θέλαμε να βελτιωθούν. Πιστεύουμε πρώτα απ' όλα ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε την καλή εφαρμογή της τωρινής οδηγίας όσον αφορά τις, χώρες, τις ώρες ανάπαυσης ενισχύοντας ε, τις κυρώσεις και τους ελέγχους. Πιστεύουμε πως δεν είναι ανάγκη να αναθεωρήσουμε το σημερινό σύστημα κατανομής ε, οδήγηση ανάπαυση έτσι όπως το προτείνει η Επιτροπή. Λειτουργούν τα συστήματα που έχουμε σήμερα και τα γνωρίζουν οι οδηγοί ούτε στη διαβούλευση που έγινε με την κοινωνία των πολιτών, ούτε κάποια άλλη στιγμή, φάνηκε να υπάρχει πρόβλημα με την περίοδο αναφοράς των δύο εβδομάδων. Γι' αυτό δεν βλέπουμε να γιατί να γίνουν τέσσερις εβδομάδες. Οι κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν τις 45 ώρες ανάπαυση ή παραπάνω να είναι εκτός φορτηγού, να μπορούν να έχουν καταλήματα οι οδηγοί και να διαλέγει το που θα περάσει την ανάπαυση αυτή που θέλει ο οδηγός. Και θα πρέπει, όπως είπα και πριν, να διασφαλίσουμε τα κατάλληλα καταλήματα και υποδομές. Θα πρέπει να θεωρείται ως χώρα του οδηγού το μέρος κατοικίας του και όχι της έδρας της επιχείρησης. Επίσης, θα πρέπει το κόστος της επιστροφής του οδηγού στη χώρα του να καλύπτεται από τον εργοδότη του. Για να βελτιωθεί η εφαρμογή των κανόνων αυτών πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ο ευφυής ταχόγραφος και να τεθεί υποχρεωτικά για να μπορεί έτσι να γίνεται καλύτερος έλεγχος όσον αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, όπως επίσης και πώς κυκλοφορεί διασυνοριακά το φορτηγό. Οπότε, εμείς προς αυτή την κατεύθυνση πάμε και υπογραμμίζω πάνω απ' όλο ότι συμπίπτουν οι απόψει μα με την γνωμοδότηση που μας παρουσιάστηκε και τι τροπολογίε του συγητή. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, η κυρία λάμπερτ. εκ μέρου των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, εκ μέρους της Καριντέλη, της ε, σκιώδουσης συγγητριά μας μιλάω. Λέει λοιπόν ότι ευχαριστεί η ομάδα μας τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έχει κάνει και η έκθεση δείχνει ότι έχουμε καταλάβει πόσο πολύ επήγει το θέμα και ότι όπως φαίνεται από την πρόταση του εισηγητή πρέπει να θέσουμε κανόνες συγκεκριμένους και αποτελεσματικούς που να μπορούν να ελέγχονται επίσης ικανοποιητικά. Συνεπώς, σας στηρίζουμε στην επιθυμία σας να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση του τομέα. Ο ψηφιακός ταχογράφος πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερα την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά θα βελτιωθεί και η ασφάλεια, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, για την ασφάλεια ολονών μας, όχι μόνο των οδηγών. Επίσης, συμφωνούμε με την διεύρυνση του πεδίου και όσον αφορά την αντικατάσταση των μεγάλων φορτηγών από ελαφρά για να αποφύγουν ακριβώς την εφαρμογή των κανόνων σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να το δούμε αυτό. Όντως θα πρέπει να είναι κάτω από 100 χιλιόμετρα μόνο η εξαίρεση. Αλλιώς όχι. Για την ανάπαυση σας είπα, όντως δεν υπάρχουν ε, ικανοποιητικά καταλήματα και υποδομές για την ανάπαυση των ε, οδηγών εκτός του φορτηγού τους πρέπει να μπορούν οι οδηγοί να επιστρέφουν στη χώρα τους ή τέλο πάντων να αποφθούν όπου εκείνοι επιθυμούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείε που αφήνουν τους οδηγούς για εβδομάδες και για μήνες στους δρόμους. Και εμείς είμαστε εδώ η Επιτροπή μας ακριβώς για να προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς από την εκμετάλλευση των εργοδοτών τους που γίνεται μερικές φορές. Άρα προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Ρώσα Νταμάτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το χρόνο οδήγηση και χρόνο ανάπαυσης των οδηγών ε, και εφόσον μιλάμε για το θέμα αυτό, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία για του εργαζομένου στον κλάδο αυτό και περισσότερη ασφάλεια και στου δρόμου. Γι' αυτό θα προσφέρω και τη δική μου συνεισφορά. Η ευθύ Σταχογράφη για να μπορούμε να καταγράψουμε σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία περιοδικών είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για να γίνονται σεβαστοί οι ημερήσιοι χρόνοι και οι εβδομαδιαίοι χρόνοι ανάπαυσης και οδήγησης. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για το κατά πόσον το εργαλείο αυτό θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Επίσης, πρέπει την ίδια σημασία να δώσουμε και στο χρόνο ανάπαυσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο, στην κατοικία του οδηγού ε, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ζώνες επαρκώς ε, ε, εξοπλισμένες όπως ασφαλείς χώρες στάθμευσης και χώροι ανάπαυσης για τους χρόνους αυτούς ακριβώς θα πρέπει οι οδηγοί να μπορούν να επιλέξουν αν θα κοιμηθούν στο όχημά τους ή αν θα χρησιμοποιήσουν ε, τους χώρους στέγασης. Θα πρέπει να γίνουν αξιοπρεπείς οι συνθήκες άσκησης του επαγγελματό τους και αυτός θα είναι και ο στόχος των τροπολογιών που θα υποβάλλονται τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε, ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το χρόνο οδηγηση και ανάπαυση των οδηγών φορτηγών, συμφωνούμε αρκετά με την πρόταση του συγητή του κ. Μπαχ. Άμα θέλετε να μειώσετε την προθεσμία για την εγκατάσταση των ψηφιακών ταχογράφων και μέχρι το 2024, που είναι μακριά ακόμα, ε, να έχουν όλα ταχογράφους ψηφιακούς και να μην υπάρχει εξαίρεση για τα ελαφρά οχήματα κάτω από 3,5 τόνους εφόσον κυκλοφορούν σε μια περιοχή κάτω από 100 χιλιόμετρα από την έδρα της επιχείρησης. Όταν θέλετε επιχειρήσεις να οργανώνουν το, την οδήγηση των οδηγών τους ώστε αυτοί να μπορούν να επιστρέφουν στο χώρο κατοικίας τους ή σε άλλο χώρο επιθυμίας τους για την εβδομαδιαία ανάπαυσή τους πάνω από 45 ώρες, δηλαδή δύο μέρες για την αντιστάθμιση μειωμένου χρόνου ανάπαυσης εβδομαδία, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης να καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού ή ανάπαυσης εβδομαδιαίας του οδηγού. Η ανάπαυση αυτή είπαμε ότι πρέπει να γίνεται εκτός φορτηγού σε ένα ξενοδοχείο δηλαδή, τέλος πάντων ή ε, στο σπίτι τους. Τέλος, χαιρετίζω την αναθεώρηση του ορισμού του χρόνου ανάπαυσης που απαγορεύει την ανάπαυση μέσα στο φωτιγό, γιατί μπορεί να συνεισφέρει να περιορίσει το μόνιμο καμποτά το οποίο σκοτώνει τις επιχειρήσεις μας και την απασχόληση στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έχω και άλλα ονόματα σε χωριστό κατάλογο. Η κυρία Λόπες Φοντανιά. Εκτός μικροφώνου, δεν την ακούμε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι ο Ζόρζο Μπάχ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ με την έκθεσή του και κυρίως με το γεγονός ότι πρέπει να προβλέπεται ένας ασφαλής χώρος ανάπαυσης με κατάλληλη, κατάλληλες υποδομές, ένα κατάλληλο κατάλημα. Σήμερα συμβαίνει αυτό μερικές φορές. Το να απαγορεύσουμε γενικά την ανάπαυση μέσα στα φορτηγά νομίζω ότι είναι υπερβολικό, κυρίως εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική για να μπορούν να αναπαυθούν εκτός Όσο δεν υπάρχουν κατάλληλε υποδομέ λοιπόν ανάπαυση, ασφαλή κτλ., δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε την ανάπαυση μέσα στο φορτηγό. Επίση, όσον αφορά την τροπολογία 4, που αναφέρονται τα ελαφρά οχήματα τα οποία δρούν ε, που είναι κάτω από 3,5 τόνους σε ακτίνα μεγαλύτερη των 100 χιλιόμετρων. Στη Σαραγώσα, για παράδειγμα, που ξέρω εγώ, επιχείρηση η οποία έχει την έδρα της μέσα στην πόλη, θα έπρεπε να μπορεί μέσα στην ίδια ε, περιφέρεια να μπορεί να δρά. Θα έπρεπε δηλαδή να αλλάξει ο αριθμός των χιλιόμετρων. Και έχω και κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τις τοπικές ή περιφερειακές εταιρείε που χρησιμοποιούν οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Κατά πόσο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία ή όχι γιατί στην περίπτωσή τους είναι και αυτές που κάνουν διεθνείς μεταφορές. Τα σου ταχογράφου όσο πιο γρήγορα τον έχουμε τόσο το καλύτερο για όλους μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Πυρίνσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του για τη γνωμοδότησή του που αποτελεί μια πολύ καλή βάση προκειμένου να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας για αυτό το θέμα. Πολύ καλά αυτά που λέει. Λοιπόν, έχω και εγώ όμως και μερικά να σημειώσω. Το πρώτο για την περίοδο αναφοράς προκειμένου να υπολογίσουμε τη την εβδομαδία συγγνώμη, ανάπαυση. Πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση του συγητή προκειμένου οι δύο εβδομάδες αντί για τις τέσσερις εβδομάδες να ισχύσουν γιατί οι δύο εβδομάδες διασφαλίζουν καλύτερα την προστασία των εργαζομένων περιορίζοντας την ευελιξία σε δύο εβδομάδες μόνο όπου μπορούν να αποφασίσουν αν θα αναπαυθούν ή όχι. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε τέσσερι εβδομάδε σαν πεδίο, περίοδο αναφορά, σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα ο οδηγό να βρει και άλλου τρόπου παραβίαση και τελικά εκμετάλλευση. Ε, που θα γίνεται από την επιχείρηση βέβαια σε βάρο του οδηγού. Χρειάζεται εκ νέου οργάνωση των ε, επιχειρήσεων ε, βέβαια τώρα έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαδρομές. Τώρα, όσον αφορά τα οχήματα τα ελαφρά κάτω των 3,5 τόνων και αν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ή όχι εδώ, δεν νομίζω ότι αιτιολογείται καλά. Δεν δικαιολογείται κατά τη γνώμη μου. Γιατί. Πώς μπορεί κανείς να κάνει διεθνείς μεταφορές με όχι όχημα 3,5 τόνων. Αν υπάρχουν ανησυχίες για παραβάσεις, ε, υπάρχουν τρόποι να περιοριστούν, χωρίς όμως να αλλάξουμε τη ρύθμιση. Τρίτο, όσον αφορά τις δαπάνες, το κόστος δηλαδή για τον οδηγό προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του και πώς θα οργανώνεται η εργασία του για να μπορεί κάθε δεύτερη εβδομάδα να επιστρέφει. Νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Έχει μια σημαντική κοινωνική διάσταση. Και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να περάσει η διάταξη αυτή, όπως προτείνει ο εισηγητής προκειμένου να επιστρέφει στο σπίτι του ο οδηγός ή να πάει κάπου αλλού εφόσον το επιθυμεί για ανάπαυση. Τέταρτο, όσον αφορά τους ευφυείς ταχογράφους. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερήσουμε την εισαγωγή των ταχογράφων αυτών. Το ότι θα κοστίσουν δεν ε, φτάνει σαν ε, επιχείρημα γιατί είναι εντελώ περιφερειακό αν το συγκρίνουμε με το κέρδος τελικά για το φορτηγό και για την επιχείρηση. Εξάλλου, πολλά σύγχρονα, τα πιο πρόσφατα δηλαδή φορτηγά, διαθέτουν τέτοιον ηλεκτρονικό ταχογράφο, οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σοντέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, δουλειά του και να του πω ότι τον υποστηρίζω σε τρία τουλάχιστον σημεία που θεωρώ ζωτική σημασία. Πρώτον, η απαγόρευση του εβδομαδιαίου χρόνου ανάπαυσης ε, στον θάλαμο του φορτηγού. Δεύτερον, η χρήση του εφιού σταχογράφου για το σύνολο των οχημάτων από το 2019 ή τέλο πάντων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ο, οι προθεσμίες που προτείνει η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα μεγάλες και βεβαίως πρέπει να καλύψουμε το νομικό κενό που υπάρχει για τα ελαφρά οχήματα. Θα πρέπει να καλύπτονται ε, από την σκοπιά των μεταφορών και θα περιορίσουμε έτσι τις καταστάσεις αθέμη του ανταγωνισμού προσφέροντας ε, περαιτέρω προστασία στους καταναλωτές. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπαχ, θέλετε να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ να τοποθετηθώ για ορισμένα θέματα, κυρία Πρόεδρε. Και πρώτα, ευχαριστώ για την αναγνώριση της προσπάθειας Νομίζω ότι για την εισαγωγή των εφιών ταχογράφων όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνει το δυνατόν συντομότερο. Για την έλλειψη χώρων σταθμεύσεως θα πρέπει να το δούμε εδώ μαζί με την έκθεση για την Ευρωβινιέτα για, τη, για τα τέλη δηλαδή που θα πληρώνονται και εκεί χρειάζεται να γίνουν, να γίνουν επενδύσεις διότι τα φορτηγά αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον αυτοκινητόδρομο παρόλο που πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να υπάρχουν ε, νυχτερινά καταλήμματα. Υπάρχει λοιπόν συνολικά πάντως ε, έλλειψη χώρων σταθμεύσεω. Γι' αυτό, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα για τους 3,5 τόνου να τα συζητήσουμε. Και θα είμαι και αρκετά εύκαμπτο ό,τι αφορά το όριο των 100 χιλιόμετρων αλλά και σε ό,τι αφορά το όριο των 3,5 τόνων, οι οποίοι 3,5 τόνοι οτιδήποτε είναι κάτω των 3,5 τόνων δεν υπάρχει στη ρύθμιση. Και αυτό οδηγεί σε αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Δηλαδή όλο και περισσότερο φορτώνουν το ίδιο φορτίο αντί σε ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο σε ένα πλήθος μικρών φορτηγών αυτοκινήτων. Και επομένως εκεί οι οδηγοί εν τέλει καταλήγουν να διανυκτερεύουν πάνω στο κάθισμα του μικρού φορτηγού αυτοκινήτου 4-5 ώρες ύπνο και μετά ξεκινούν και πάλι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι περιθωριακό ή είναι μικρός ο αριθμός. Όχι. Προχωρεί πολύ αυτό το business model και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Και εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να μπορούμε να το προλαμβάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή να, να, βλέπουμε και μπροστά. Η παρούσα ρύθμιση για την ανάπαυση εκτός θαλάμου του φορτηγού ή και εντός εφόσον είναι περιορισμένη η περίοδος αναπαύσεως θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και μέσα στην καμπίνα του φορτηγού. Είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό η παρατεταμένη περίοδος αναπαύσεως ή μάλλον το πω αλλιώς, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις έχει ενδιαφέρον η πρόταση της Κομισιόν κατά το ότι η αποζημίωση που προτείνεται στον οδηγό συνδυάζεται με παρατεταμένη περίοδο αναπαύσεως σε κατάλληλο κατάλημα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να δεσμευτούμε για το αν θα είναι 2, 3, 4 εβδομάδες. Θα πρέπει οι εξαιρετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν ε, να συνοψιστούν κάπου και να υποστηριχθεί η πρόταση της Κομισιόν εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ αγαπητέ Μπαχ. Μήπως η Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι τι. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω η συζήτηση ήταν ε, πρόσφορη και πολύ επικοδομητική δείχνει το πόσο αλληλένδετη είναι οι διάφοροι φάκελοι, τα θέματα αυτά της κυρίας Λόπε Φοντάνια, της κυρίας Ενάλοβα και του κυρίου Μπαχ. Όπως ξέρετε, ο τομέας των οδικών μεταφορών είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία με 5 εκατομμύρια εργαζομένους τουλάχιστον και ορίζουμε την πρόταση να υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις και καλύτερη λειτουργία του τομέα αυτού, καθώς και ίση κανόνες παιχνιδιού, δίκαιος ανταγωνισμό. Έχουμε επίσης κατά νου ότι καλό θα ήταν να μειωθεί και το, και το διοικητικός φόρτος για τις μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να, να επιζητήσουμε υλοποίηση με πολύ σαφείς κανόνες. Η συζήτηση ε, ε, διεξάγεται αυτή τη στιγμή και στην Επιτροπή Τραν και καλό είναι να έχουμε υπόψη ότι αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Έχουν να κάνουν από τη μια με την πρόσβαση στην αγορά και την απόσπαση και από την άλλη τη διασφάλιση ε, νόμιμου ανταγωνισμού για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει τα επαγγέλματα αυτά να γίνουν ελκυστικότερα γιατί πρέπει ε, να ε, φροντίσουμε και για την κατάσταση των ε, αυτοκινητοδρόμους, να δούμε τα τέλη κυκλοφορίας, να οικοδομήσουμε, να πάρουμε πάνω τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας και να οικοδομήσουμε χώρους στάθμευσης, όπου μπορούν, μπορούν να αναπαυθούν πραγματικά οι οδηγοί. Και θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε τις εικονικές εταιρείες, τις εταιρείες γραμματοκιβώτια, καθώς και να προωθήσουμε την χρήση των ταχογράφων Χρειαζόμαστε απλούς κανόνες εύκολους να εφαρμοστούν και αυτό με οδηγεί ε, στην ε, έκθεση της κυρίας Τζαμπάλοβα η οποία είναι σημαντική γιατί θέλουμε να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες που θα ισχύουν στον τομέα αυτό τον ειδικότερο με τους κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζουμε την άποψη που πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την απόσπαση των οδηγών οδηγών που εργάζονται στο τομέα των μεταφορών δηλαδή και αυτό σε μεγάλο μέρος είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσει καλά το σύστημα. Καλωσορίζουμε τις απόψεις που εκφράζονται στην έκθεση. Οι κανόνες περί απόσπασης πρέπει να ισχύσουν και για τις δράσει καμποτάζ, διότι πρόκειται για εγχώριες δράσεις και δεν πρέπει να ισχύουν σε περίπτωση διέλευσης θα πρέπει να το δούμε αυτό σε επίπεδο διεθνών μεταφορών επίσης, Θα τα συζητήσουμε κι άλλα και Και όντω θα πρέπει να φροντίσουμε να μην εφαρμόσουμε του ίδιου κανόνε μακροχρόνια απόσπαση για την περίπτωση οδήγηση. Η μακροχρόνια απόσπαση σημαίνει συνέχεια παροχή τη υπηρεσία από τον εργαζόμενο σε κράτο υποδοχή. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για του οδηγού στον τομέα των μεταφορών ακριβώ. Γι' αυτό καλό να υπάρχει εδώ μια συγκεκριμένη μνήμα που να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Τέλο για το διοικητικό άκτο συνολικά. Νομίζουμε ότι και καλό είναι και θετικό κάποιοι από τους ελέγχους να πάνε από το σκέλος των δρόμων και τις υποχρεώσει του οδηγού στους ελέγχους στον ε, τόπο που εδρεύει η εταιρεία που απασχολεί τους εργαζομένους και να υπάρχουν εφόσον ε, γίνεται δηλώσεις σε τυποποιημένα έντυπα. Αυτά θα ε, απλοποιήσουν τη δουλειά των οδηγών. δεν είναι η βασική του δουλειά να καλύπτουν διοικητικέ υποχρεώσει. Καλωσορίζω και την έκθεση του κυρίου Μπαχ. Ιδίω τι απόψει του για την επιβολή των κανόνων και τη ε, αξιοπρεπή συνθήκη εργασία ώστε να αποφύγουμε τη στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Ακόμη και αν δεν είχε προταθεί από την Επιτροπή, ε, καλωσορίζουμε τους κανόνες για την όσο το δυνατόν εγκαιρότερη χρήση των ταχογράφων. Συμφωνούμε εδώ και προτείνει ο κύριος Μπάχ ότι θα πρέπει να είναι το 2024 να σας ενημερώσω ότι στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή διεξαγάγεται μελέτη για, την τεχνα... για το κατά πόσο θα είναι τεχνικά εφικτό κάτι τέτοιο καθώς και για τον εξοπλισμό των φορτηγών ποιο θα είναι το κόστος. Υπάρχουν φορτηγά με φύς που θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς στο μέλλον ήδη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα πάρουμε παράδειγμα και να δούμε ότι είναι ρεαλιστικό όταν λέμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάντω σίγουρα θα είναι μια ημερομηνία κοντινή σε αυτό που πρότεινε ο κ. Μπαχ. Απλώ περιμένουμε να συγκεντρώσουμε και τα απαραίτητα στοιχεία για να το υποστηρίξουμε. Σημειώνω την γνωμοδότηση για την άποψη για τα ελαφρά εμπορικά ε, οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Πρόκειται για μια τάση που αναδύεται το Λένα και ισχυρότερη. Υπάρχουν κάποιε εξελίξει που οδηγούν προ τα εκεί. Είναι όμω νωρί για να δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτή η τάση, αυτή η δυναμική πρόθεση της Επιτροπής στην πρότασή της ήταν να προτείνει τα πρώτα βήματα για την επαγγελματική μεταχείριση του κλάδου των οδηγών αυτών των ελαφρών φορτηγών. Έχουμε επίσης κάποιες αμφιβολίες περί αναλογικότητας για το κατά πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε τις ίδιες υποχρεώσεις περί ταχογράφων στις εγχώριες δραστηριότητες και πρέπει να σας ενημερώσω ότι σε, άλλα, σε άλλες περιπτώσεις ε, συζητιέται το όλο θέμα αυτό από την άποψη των διεθνών κανόνων για τα βανάκια. Ο κύριος Μπαχ έχει εισάγει την έννοια της ακτίνας των 100 χιλιόμετρων. Ε, 100 χιλιόμετρα λοιπόν, αλλά για διεθνείς μεταφορές και όχι εγχώριες και μετά να δούμε αν θα ισχύει ε, συνολικά το σύστημα των κανόνων ή όχι. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για έναν τομέα στον οποίο δεν θέλουμε να επιβάλλουμε διοικητικό άχθο, διότι μιλάμε για τομέα με πολλέ μικρομεσαίε κυρίω, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει με τα βαρέα φορτηγά. Χαίρομαι πολύ που ο συγκεκριτή προτείνει κανόνε για την ε, αποζημίωση και το τι πρέπει να ισχύει για την ημερήσια ανάπαυση σε, σε αντιδιαστολή με την εβδομαδιαία ανάπαυση. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά και θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλο έλεγχο. Επίση και για σκοπού οδική ασφάλεια. Σημαντικό είναι η αρχή ότι ο οδηγό θα πρέπει συστηματικά να επιστρέφει σπίτι του. η κατοικία του ή άλλος χώρος ιδιωτικού ε, χαρακτήρα όπως πολύ συχνά προκύπτει και από τους ορισμού της Επιτροπής. Δεν θέλω τώρα να επανέλθω στο τι θα εννοήσουμε με το συστηματικά, τρει, τέσσερι πέντε εβδομάδες, τέλος πάντων μία μηνιαία επιστροφή στο σπίτι. Για να μην καταντήσουμε να έχουμε μόνο ομάδες οδηγούς πλανόδιους εντελώς. Ε, και τελευταίο, εξίσου σοβαρό, δεν αναφέρθηκε στη συζήτησή σας, αλλά το θεωρώ σημαντικό, η τροπολογία 12 στην έκθεση του κυρίου Μπαχ, η οποία αναφέρεται στην αποζημίωση βάση των επιδόσεων των οδηγών. Θέλω να γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτή τη στιγμή τον υπολογιστή αποζημίωση των οδηγών. Με μια απλή απαγόρευση μπορεί να έχουμε ανεπιθύμητες συνέπειες για το επίπεδο των αποζημιώσεων των οδηγών. Η Επιτροπή την τροποποίησε την πρόταση αυτή και λέει ότι αυτό επιτρέπεται όπου δεν ε, μπαίνει σε κίνδυνο η ασφάλεια των αυτοκινητοδρόμων. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιο είναι το σωστό επίπεδο αλλαγής για την πρόταση της Επιτροπής. Κατά την κατανόησή μου, η διάταξη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνει τον εργοδότη του οδηγού να προσφέρει στέγη, να καλύψει το κόστος της στέγης. Κάτι που νομίζω ότι το προβλέπει και η πρότασή του εισηγητή. Ευχαριστώ. Thank you. That means that we... Ευχαριστούμε. Καθώς προχωρούμε στην τρίτη σχετική έκθεση μέσα από το ίδιο σύνολο Μιλάμε για την τροποποίηση κανονισμών για να προσαρμοστούν στις εξελίξεις του κλάδου. Να δώσω το λόγο στην κυρία Λόπε Φοντανιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντως και η έκθεση αυτή, η τρίτη γνωμοδότηση δηλαδή, δεν είναι πολύ καλά με τις δύο προηγούμενες. Ακούσαμε εξετάζοντας τις δύο προηγούμενες, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, συχνά. Το ίδιο προφανώς ισχύει και με τη δικιά μου γνωμοδότηση, το ξέρω από τις συναντήσεις που είχαμε με τους σκιώδεις. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες και είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών και να τηρήσουμε βέβαια και κάποιες ρυθμίσεις ασφάλειας αλλά και εργασιακές. Στι διάφορε χώρε, ακόμα και μεταξύ των διαφόρων εταιριών υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Αλλά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Είναι βασικό αυτό και πολύ καλό για τον κλάδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, ποια είναι τα σημεία που θέλω να υπογραμμίσω. Είναι τα εξή. Πρώτον, δεν πρέπει να δημιουργούνται υπερβολικά διοικητικά εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοπασχολούμενους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν έχουμε αρκετούς οδηγούς. Οπότε δεν πρέπει να επιβάλλουμε υπερβολικούς περιορισμούς σε αυτούς που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα. με τις δυσκολίες που βάζουμε στις εσωτερικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πλήξει και την ε, οικονομία μας. Οι μεταφορές προσφέρουν απασχόληση και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Κυρίως για τους οδηγούς ε, ελαφρών ε, φορτηγών κάτω των 3,5 τόνων. Από την άλλη, δεν πιστεύω ότι θα ήταν καλό η οδηγία για τους αποσπασμένους να χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας. Τουλάχιστον όχι έτσι όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κανόνες καλύτερα προσαρμοσμένη στον κλάδο. Όσον αφορά το καμποτάζ, το καμποτάζ έχει σαν στόχο να εμποδίσει την επιστροφή με κενό το φορτηγό. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια αποδοτικότητα γιατί αλλιώς όπως ε, καταλαβαίνετε θα αυξηθεί πολύ το κόστος μεταφοράς. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να συμπεριληφθεί, να μην συμπεριληφθεί το καμποτάζ στην οδηγία για τους αποσπασμένους. Αν αποφασίσει η πλειοψηφία να συμπεριληφθεί, τότε θα έπρεπε να πετύχουμε συμφωνία για να διευρυνθεί ο αριθμός των ημερών που επιτρέπεται για την επιστροφή στη χώρα του οδηγού. Αυτό που πρέπει να εγγυθούμε είναι την επιστροφή στη χώρα μέλος, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία και να μην γίνονται εθνικές μεταφορές σε τρίτη χώρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι έλεγχοι. Ανάμεσα στα επιχειρήματα που ακούγονται για την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους ακούγεται το κοινωνικό ντάμπικ, οι κακές συνθήκες εργασίας των οδηγών ή η έλλειψη εργασιακής ασφάλειας για τους οδηγούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές και εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε. Αλλά δεν ισχύει στις περισσότερες ε, εταιρίες διεθνών μεταφορών, οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ισχύει παντού, σε ολόκληρο το τομέα. Πάντα είμαστε υπέρ της διαφοροποίησης ε, προσφοράς υπηρεσιών, εγκατάστασης, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στην ενιαία αγορά. Συγχρόνως όμως η ελευθερία εγκατάστασης πρέπει να σημαίνει πραγματική παρουσία στη χώρα. Άρα πρέπει να γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και πιο πολυάριθμοι που να διασφαλίζουν αυτή την πραγματική παρουσία στην χώρα που έχει την έδρα της η επιχείρηση και έτσι να καταπολεμήσουμε τις εικονικές επιχειρήσεις. Μιλάμε επίσης και για τους ευφύς ταχογράφους. Και αυτό για να καταπολεμήσουμε τις εικονικές επιχειρήσεις και να γίνεται καλύτερος έλεγχος. Πιστεύω και εγώ ότι είναι κάτι σημαντικό και συμφωνώ με αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Uh, I'll give the Ευχαριστούμε. Ο Σον Σάιμον έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ, καθώς και τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έχει κάνει, καθώς και τους άλλους κοιόδης εισηγητάς για την επικοδομητική τους προσέγγιση. Το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητού περιλαμβάνει 24 τροπολογίες, ορισμένες από τις οποίες μας βρίσκουν σύμφωνους αύξηση δηλαδή των προτινόμενων ελέγχων συμπόρφωσης, αντιμετώπιση του θέματος των ε, εταιριών χρηματο, ε, γραμματοκιβωτίου. Ορισμένες άλλες θα είναι πιο δύσκολο να τι υποστηρίξουμε, όπως για παράδειγμα είπε οι τροπολογίε που αναφέρονται στην ε, ε, απόσπαση για καμποτάζ. Όμως είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι όπως είπε η ίδια η Μαρτίνα και κατ' επανάληψη μάλιστα, όλοι έχουμε συμφωνήσει στις ανεπίσημες συζητήσεις μας των σκιωδών ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες που πραγματικά να αποδίδουν και να μπορούν να εφαρμόζονται και να είναι ρεαλιστική η διαδικασία και η προσέγγιση χωρίς ιδεολειψίες ή θεωρητικολογίες. Σύντομα τώρα για κάποιες από τις τροπολογίες του εισηγητού και πάλι σύντομα μετά σχετικά με ορισμένες δικές μας. Για τις ε, εταιρείε γραμματοκιβωτίου συμφωνεί, συμφωνεί ο εισηγητής και χαίρομαι γι' αυτό. Τροπολογίες 5 και 6 λέει να πάψουν αυτές οι επιχειρήσεις να καλύπτουν βέβαια αυτοαπασχολούμενους. Το ίδιο και για τα ελαφρά οχήματα που σύμφωνα με την πρόταση της ε, Επιτροπής συμμορφώνονται με δύο από τα τέσσερα κριτήρια πραγματική εγκατάσταση και οικονομική απόδοση. Αντίθετα με, τις, ε, με την τροπολογία 30 της συγκητρίας θεωρούμε ότι τα οχήματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στα τέσσερα κριτήρια. Επομένως και επαγγελματική ε, απόδοση κλπ διότι είναι και το, το τμήμα εκείνο της αγοράς όπου σημειώνονται οι περισσότερες παραβιάσεις. Επομένως φαίνεται λάθος να αποκλείσουμε το τμήμα αυτό της αγοράς από τα μισά κριτήρια. Είναι μεν αληθές ότι η μελέτη δικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει και ένα κόστος συμμόρφωσης, αυτό όμως δεν εξαντλεί το θέμα, διότι η μελέτη δικτύπου επίσης προβλέπει εξοικονομήσεις στον τομέα Τη τάξη των 2,7 έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα υπάρχει αντάλλαγμα. Τώρα για τι απαιτήσει οικονομικής δυναμικότητας, η τροπολογία 18, η συγκίτρια προτείνει διαφορετικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μικρότερα φορτηγά. Διαρωτώ με όμως από πού προέρχονται οι αριθμοί που ε, προβάλλει τα χίλια ευρώ για παράδειγμα δεν είναι σαφές για την απόσπαση 7, 16, 21 και 22 τροπολογία λυπούμεθα που η συγκέντρια προτείνει να βγει η απόσπαση από το καμποτάζ εμείς προτείνουμε να μπει το καμποτάζ στις ρυθμίσεις αυτές, διότι θεωρούμε ότι συνδέεται άμεσα. Για τους ελέγχους και για την επιβολή των ρυθμίσεων όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η συμμόρφωση και γι' αυτό υποστηρίζουμε άλλωστε την τροπολογία 23 για την αύξηση των ελέγχων, αν και θα πρέπει να φανούμε πιο φιλόδοξοι. Για τις δικές μας τροπολογίες όταν θα τις καταθέσουμε θα πω το εξής. Ναι, πρέπει να επιμείνουμε στην ε, προσωρινή φύση του καμποτάζ, αλλά και στην ελευθερία εγκατάσταση των εργαζομένων. Και είτε θα πρέπει να περιοριστεί η περίοδος του καμποτάζ, όσο δεν ισχύει η νομοθετική ρύθμιση για τις αμοιβέ ή θα πρέπει ίσως να μείνουμε κάπου κοντά στους ισχύοντες κανόνες, να μην αλλάξουν πολύ. Τα έγγραφα να παραμένουν στο αυτοκίνητο για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης. Να εγκριθεί και ε, το, η ηλεκτρονική φορτωτική και δεν θεωρούμε ότι η εισαγωγή του εφιού σταχογράφου μέχρι το 2024 είναι πραγματικά ταχεία. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον αργή και θα θέλαμε ο ηλεκτρονικός ταχογράφος να αρχίσει να μπαίνει, να αρχίσει να ισχύει τέλο πάντων από το τέλος του 2021 και αναμένουμε και στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν αυτό είναι εφικτό και αν όχι γιατί όχι. Επίσης το ηλεκτρονικό μητρό των επιχειρήσεων, το Social Guarantee Fund για την οικονομική δυναμικότητα. Να υπάρχουν λοιπόν, χρήματα για για την κάλυψη αποζημιώσεων για ε, ζητήματα υγείας, ε, απολύσεις κλπ. Και εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Σον. Η κυρία Στίβενς. Ορίστε κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της που όντως εκφράζει την επιθυμία να αντιμετωπιστούν οι εικονικές επιχειρήσεις, οι ψευδοαπασχολούμενοι κλπ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να παίζουν ένα σωστό παιχνίδι, δίκαιο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σκληρύνει τους κανόνες. Και αυτό είναι θετικό. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο οι απαιτήσει που προτείνει η Επιτροπή είναι κατάλληλες και είναι παρκείς. Εγώ αμφιβάλλω. Πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να είναι παρόν κάποιος από την επιχείρηση εκεί που βρίσκονται οι δραστηριότητες, δεν ξέρω αν είναι το σωστό. Όσον αφορά το καμποτάζ, Πάλι στηρίζω την εισηγήτρια ότι οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, αλλά πρέπει να είναι και εφαρμόσιμοι, ρεαλιστικοί. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να καταργήσει κάποια ανώτατα επίπεδα. Γιατί έτσι κι είναι δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση και άρα ε, υπάρχει περίπτωση να γίνουν ε, απάτες. Έπειτα, το περιβάλλον είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να υπάρξει κάτι και γι' αυτό. Όμως μια μικρή χώρα σαν τη δικιά μου μπορεί με 5-7 μέρες να κάνει πολύ περισσότερα. Είναι γεγονός ότι το καμποτάζ δεν πρέπει να βοηθήσει για να γίνονται περισσότερες ε, απάτες. Πάντως εγώ εύχομαι στην εισηγήτρια να έχει μια όσο γίνεται καλύτερη γνωμοδότηση στο τέλος. Thank you. Then I'll give the floor to, uh, Ευχαριστούμε κυρία Τζαμπάλοβα. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική. Καλωσορίζω την έκθεση της κυρίας Λόπε Φοντανιέ. Διότι έχετε λάβει υπόψη αυτό που χρειάζεται ε, περισσότερο αυτή τη στιγμή. Μια συνολική έποψη. Το αναφέρετε και στο σχέδιο γνωμοδότησής σας τα διαφορετικά θέματα που συζητιούνται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πρέπει να συμβαδίσουν. Είναι αλληλένδετα, αλληλοσχετίζονται. Απόσπαση εργαζομένων, απόσπαση οδηγών. Ο δικός, ε, το δικό σα θέμα έχετε συμπληρώσει όλη την εικόνα. Πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να δούμε το κόστος του καμποτάζ, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς... τη μείωση του διοικητικού άχθου, το να αποφύγουμε το διοικητικό φορτό, την κατάσταση των μικρομεσαίων στον τομέα των μεταφορών και την ανάγκη να υπογραμμίσουμε πόσο απαραίτητη είναι η έλεγχη. Πρέπει νομίζω να πούμε από τώρα ότι προβλέπουμε ε, αρμονική συνεργασία στις συνεδρίες των σκιωδών και σίγουρα ο οδηγός μεταφορών λόγω της ε, φορητότητάς του του γεγονότος ότι βασίζεται στην κυκλοφορία χρειάζεται δική νομοθεσία. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρόνια Κάρη από την GUNGL έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τέτοιον καλό διάλογο σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Πάνω απ' όλα ε, βεβαιωνόμαστε, ε, πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι έχουν νόμιμες αποζημιώσεις οι οδηγοί μας. Ε, πριν από λίγες μέρες είχα τηλεφώνημα από τον δανεικό οργανισμό που ασχολείται με εργαζόμενους από διαφορετικές χώρες και καταγράφει τα στοιχεία τους, τους πληρώνει με τις δικές μας αμοιβές, με το δικό μας επίπεδο αμοιβών. Και ο οργανισμός μας ε, ε, ξέφρασε την απογοήτευσή του και την ε, αγανάκτησή του, διότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από μεγάλες εταιρείες, από πολλές εταιρείες μάλιστα, που πιέζουν για να εφαρμόσουν χαμηλότερες αμοιβέ. Να προσφέρουν χαμηλότερες αμοιβέ, κάνοντας αθέμητο ανταγωνισμό προς τις μικρότερες. Εκεί λοιπόν πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός και ίσοι κανόνες παιχνιδιού για όλους. Το πρόβλημα αρχίζει με το κατά πόσον οι οδηγοί μπορεί να παραμείνουν πολλές μέρες κάπου πριν ξεκινήσουν το καμποτάζ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυστηρότερους κανόνες. Εδώ, στην ομάδα μου, Θεωρούμε ότι το καμποτάζ μπορεί να γίνει ε, μετά από ένα ταξίδι πολλών ημερών και την παραμονή σε μια χώρα, δηλαδή με τη χώρα προέλευσης και ένα επόμενο κράτος να ε, καταγράφουν τα στοιχεία. Απλώς θα μπορούσαμε να ε, επιτρέπουμε μία περίπτωση καμποτάζ ανά ταξίδι. Ιδάλω, αν αυτά συσσωρεύονται σε σχέση με του ντόπιου οδηγού ενό κράτου μέλου, αρχίζει να υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Επίση, για το χρόνο ανάπαυση. Αν κάποιο έχει ε, κάνει καμποτάζ, πρέπει να φύγει από τη χώρα πριν επιστρέψει για να ξανακάνει καμποτάζ. Αυτό είναι ίσως η διαφορά σε σχέση με τους κανόνες περί απόσπασης. Ένας από τους τομείς όπου συμφωνούμε περισσότερο με την πρότασή σας είναι στα αποτελέσματα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι έχετε μια σειρά από προτάσεις για να καταπολεμήσετε τις εικονικές εταιρείε, τις ε, εταιρείε που βασίζονται σε γραμματοθυρίδες. τα ταχυδρομικές θηρίδες μόνο. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να καλύπτονται περισσότερα οχήματα και όχι λιγότερα. Εδώ λοιπόν ε, η πρόταση για το, όρος, για το όριο στο βάρος θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Σήμερα είναι πολλές οι εταιρείε που χρησιμοποιούν ακριβώς τα μικρότερα οχήματα, τα βανάκια, για να διαφεύγουν από τους κανόνες. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε να μην υπάρχει απλώς μια παράκαμψη των κανόνων και να κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι με διαφορετικά οχήματα. Αναμένουμε στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε. Εκπροσωπεί κανείς τους πρασίνους. Α, κανείς δεν έμεινε. Η ευθυντή. Κανείς ούτε από εκεί. Ο κύριος Μαρτά, η ΕΝΕΦ, έχετε το λόγο. Όχι. Δεν θέλετε. Πάμε στον κατάλογο αγορτών. Η κυρία Σαντέρ έχει το λόγο. Σαντέρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λόπε Φουντανιέ για τη δουλειά που έχει κάνει ήδη και όσα θα κάνει και στη συνέχεια. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολα. Συμφωνώ. Συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν λέει ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε πρακτικές αθέμητες, ιδίω όταν αναφέρει τη μάστικα των εικονικών εταιριών, ταχυδρομικών θηρίδων. Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι έλεγχοι και αποτελεσματικές κυρώσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φανταστούμε σκεφτούμε, να σκεφτούμε προτάσεις για να προβλεφθούν κριτήρια ώστε να μπορεί κανείς να πιστοποιεί μια δραστηριότητα, πραγματική δραστηριότητα στη χώρα προέλευσης, ίσως κριτήρια κύκλου εργασιών ε, με την αρχή που εφαρμόσαμε και για την περίπτωση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλειας με τις τροπολογίες που Απέναντίας για το θέμα του καμποτάζ η θέση μου διαφέρει προφανώς. Οι συνθήκες της απόσπασης πρέπει να εφαρμόζονται από την πρώτη μέρα. Και πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε ένα τότατο όριο για τις δραστηριότητες που θα επιτρέπονται. Το καμποτάζ είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Για να μην γυρνάει άδειο το φορτηγό. Αλλά μην ανοίγουμε την πόρτα στον αθέμητο ανταγωνισμό με τους ντόπιου οδηγούς. Ευχαριστώ. Thank you, Madame Sander. Now it's uh, Mr. Pirinski. The floor is yours. Ευχαριστούμε κυρία Σαντέρ. Ο κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Θαυμάσιο το έργο της συζητήτριας. Θα σύντομος. Η απέτηση για την πραγματική εγκατάσταση. Χαίρομαι που τίθεται το θέμα αυτό. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη την ανάγκη της επιβολής πραγματικών ελέγχων στις επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών. διότι χρειάζονται έλεγχοι για τις επιχειρήσεις αυτές, διοικητικοί, και είναι αναγκαίο να τονιστεί η πραγματική εγκατάσταση, πραγματική έδρα δηλαδή, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τώρα, για την συμπερίληψη των ελαφρότερων φορτηγών. Εδώ υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Συμφωνώ με τα όσα είπε προηγουμένως ο Σον Σάιμον. Την αποφυγή δηλαδή της κατάχρησης των οχημάτων αυτών. Όμως υπάρχουν και θέματα πρόσβαση στην αγορά των μικρότερων επιχειρήσεων. Όταν αυτές σέβονται και συμμορφώνονται με τους υφιστάμενους κανόνες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα εδώ και επομένως η ανάγκη νομίζω να σχολιάσει και η Επιτροπή με την έννοια δηλαδή να σχολιάσει για τα μικρότερα φορτηγά αυτοκίνητα για να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην αποφυγή της χρήσης των αυτοκινήτων αυτών χωρίς από την άλλη μεριά να παρεμποδίζονται οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις από το να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Τώρα για την ίδια την φύση του καμποτάζ που είναι προσωρινή και όχι διαρκή σε δραστηριότητα και την αποφυγή του παράνομου καμποτάζ η πρόταση αξίζει να υποστηριχτεί Χρειάζεται βέβαια προσεκτική προσέγγιση, διότι οι ενδεχόμενες παραβιάσεις θα είναι διοικητικού χαρακτήρα και όχι ποινικού. Με την επιβολή επομένως κυρώσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ναι. πρόσοχη ώστε να μην φυγούν υπέρμετρα τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την περίοδο για την απέτηση της εφαρμογής των κανόνων της απόσπασης, αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι αυτό είναι ορθό, θα είναι σωστό να διατηρηθεί η περίοδος των 7 ημερών και όχι των 5 ημερών προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ληφθεί υπόψη και η άρση της επιβολής των μειωμένων ημερών καμποτάζ. Και τέλος, για τους κανόνες, για την επιβολή μάλλον των κανόνων, είναι αναγκαίο να είναι αποτελεσματική έλεγχη αυτή. Ο διπλασιασμός του ελάχιστου αριθμού δειγματοληπτικών ελέγχων σε σύγκριση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι σωστό αυτό, δηλαδή προτείνει η συγγήτρια. Θα σημάνει ένα έξτρα, βάρο, ένα έξτρα βάρος για τα ελεγκτικά όργανα που είναι όμως δικαιολογημένο εν ώψη των αποτελεσμάτων που επιδιώκουμε. Okay, thank you. Ωραία, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου συζητήσαμε τρεις διαφορετικές εκθέσεις. Προφανώς και είναι σαφές μετά από τη συζήτηση έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. και για το χρονοδιάγραμμα. Έχουν παρόμοιο χρονοδιάγραμμα. Υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 30 Ιανουαρίου το μεσημέρι στις 12. Εξέταση των τροπολογιών εδώ στις 26 και 27 Φεβρουαρίου. Έγκριση στην Ολομέλεια 25 5 28 Μαρτίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών στις 15 Μαΐου και έγκριση στην Ολομέλεια αρχές καλοκαιριού ή τέλος πάντων ε, τέλος άνοιξης. Αυτό για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ όλους για την ε, παρουσία τους. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας άκουσε και να θυμίσω ότι θα αρχίσουμε στις 2.30, 14.30 το απόγευμα. Ε, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει. με την υποδοχή της νέας Προεδρίας, τον Προεδρεύοντα, τον κύριο Παϊκόφ, ο οποίος είναι Βούλγαρος ε, Υπουργός ε, Απασχόλησης. Παρακαλώ να είστε εδώ παρούσες και παρόντες, διότι από τις συζητήσεις που είχαμε τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κατά τη Βουλγαρική Προεδρία θα περάσουν πολλά σημαντικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει την Επιτροπή μας και ε, επηρεάζουν όσα έχουμε κάνει και όσα θα κάνουμε εδώ να είστε στην ώρα σας. Δυόμιση. Όταν θα έρθει ο κύριος Βέκοφ. Να πω ότι είχαμε και το πέμπτο, τον πέμπτο τριμερή διάλογο για την απόσπαση των εργαζομένων. χθες το βράδυ. Όλη τη νύχτα. Πολύ μεγάλη στιγμή για μας. Και πολύ καλή για να συναντήσουμε τον Υπουργό Εργασίας θα σας δω σε λίγο. Θα υπάρχει διερμηνία στα βουλγαρικά. Θα έχουμε διερμηνία στα βουλγαρικά. Ναι, μα το Θεό. Thank you and see you soon again. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αργότερα.